Uh, well, good afternoon, everybody. And a very warm welcome to our... Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην σημερινή μας ε, ακρόαση ε, που αφορά την εσωτερική αγορά υπηρεσιών, περιγραφή της κατάστασης και επόμενα βήματα. Όπως έτσι δεν είναι η αρχική διατύπωση, αλλά έχει ενταχθεί και στο πρόγραμμα της Επιτροπής ε, για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Θα έχουμε λοιπόν μια σημαντική συζήτηση σήμερα το απόγευμα για το πώς ε, η αγορά, η οδηγία περί υπηρεσιών θα μπορούσε ε, να συμβάλλει και κατά πόσο συμβάλλει ή όχι και τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Να καλωσορίσω θερμά όλους τους ομιλητές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ έχουν λάβει οδηγίες για τον χρόνο ομιλίας. Γενικά έχουμε ένα ρολόι πολύ φιλικό προς το χρήστη, το οποίο θα ε, παρουσιάζεται μπροστά σας για να έχετε και μια αίσθηση του χρόνου. Να καλωσορίσω και τα μέλη του Κοινοβουλίου και όσους ενδεχομένως ε, παρακολουθούν ε, μέσω web stream ακρόαση εντάσσεται ε, στις εργασίες ε, που έχει αναλάβει ε, η συγγήτρια Άννα Μαρία Κορέσα Μπίλτ με έκθεση πρωτοβουλίας. πολύ σύντομα θα της δώσω το λόγο για να παρουσιάσει το θέμα και θα εστιαστούμε Πρώτον, στην ανταπόκριση στην ε, κρίση, άρση εμποδίων και απελευθέρωση των ε, υπηρεσιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη. Και δεύτερον, κατά πόσο παρακολουθούμε την καινοτομία και μεγιστοποιούμε τα ωφέλη για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Και έχουμε και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ε, παρουσιάσεις για το πώς μπορούμε να σωματώσουμε και την πληροφορική σε αυτόν τον τομέα αλλά και τις πτυχές που αφορούν τους καταναλωτές σε ό,τι αφορά την οδηγία περί υπηρεσιών. Γιατί βεβαίως βοηθάμε έτσι και τους καταναλωτές να αντιμετωπίσουν ζητήματα που έχουν σχέση με την πρόσβαση ε, στην αγορά και στις υπηρεσίες. Να παρουσιάσω εν συντομία τους ομιλητές πριν περάσουμε στα επόμενα ζητήματα. Όμως θα έχετε λάβει κι εσείς ε, κάποια έγγραφα με το βιογραφικό σημείωμα των ε, ομιλητών. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Να καλέσω λοιπόν την εισηγήτρια. Αναμαρία Κόρα Μπίλτ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές που έχουν ταξιδέψει από μακριά για να έρθουν σήμερα εδώ και όσους μας ακούν από το σπίτι. Οι καλέ ειδήσει είναι ότι ο Μάρτιν δεν είναι μόνο ο Πρόεδρος, αλλά και σκιώδης από πλευρά ACR. Και ε, είχαμε και άλλους εξαιρετικούς ε, σκιώδης ε, εισηγητές, όπως η κυρία Ράπτη που φτάνει τώρα, κύριος Λόκεγκάρτ από, από την Άλντε, κυρία Ρούλερ από τους Πρασίνους. Και βλέπω και τον κύριο Γκέπερντ με τα χαράς που έχει μια, αναλάβει μια αντίστοιχη έκθεση και την κυρία Μικροζάντα που θα μας ε, συνοδεύσει. Το συζητούμε αυτό το θέμα από το 2006 πλέον. Και είχαμε την προθεσμία υλοποίηση ε, του 2009 και παρόλα αυτά πολλά κράτη-μέλη δεν την έχουν υλοποιήσει. Ο κίνδυνο τώρα, μπορείτε να διαβάσετε και το άρθρο, σας συνιστώ να το κάνετε, γιατί παρουσιάζει κάποιες από τις κατευθυντήριες γραμμές ε, ε, που έχουμε παρουσιάσει στις επιτροπές και έχουν ε, πολύ ισχυρή εντολή για την μη ανοχή σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, που συνάδει και με τις απόψεις του κυρίου Μπαρνιέ. Κάποιοι λένε, και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ίσω είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι. Ίσως ε, οι προσδοκίε να ήταν ε, υπερβολικά αυξημένε σω να μην υπάρχει τέτοια δυναμική εδώ. Εγώ λέω όχι, λάθο, Δεν πρέπει να επικεντρωθούμε στην ε, οδηγία περιπηρεσιών, αλλά στην υλοποίηση των πλευρά κρατών μελών. Πού είναι η Ελληνική Προεδρία, εσεί πρέπει να αναλάβετε αυτό το δύσκολο έργο, αλλά προσβλέπουμε σε έναν επικοδοματικό διάλογο μαζί σα για να γνωρίζουμε περισσότερο για το τι κάνουν τα κράτη-μέλη, πώ αιτιολογείται ενώπιον των Ευρωπαίων πολιτών το γεγονός ότι ένας από τους βασικούς τομείς που έχει πραγματικές, ε, πραγματική δυναμική για την ε, ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασία ε, με τομέας που δεν ε, ε, επηρεάζει αρνητικά το δημόσιο χρέο. Πώς εξηγείτε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν θάσει τις θέσει εργασία τους, εσείς παρόλα αυτά δεν έχετε καταφέρει να άρετε τα εμπόδια και τις δυσκολίες μετά από τόσα χρόνια. Η δική μα δουλειά σήμερα λοιπόν είναι να βρούμε την προστιθέμενη αξία μετά από όλη τη δουλειά που έχει γίνει. Το επίκεντρο λοιπόν σήμερα είναι το εξή. Πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερε θέσει εργασία. Όχι ποιε είναι οι εργασίε, οι συνθήκε εργασία μάλλον. Έτσι κι αλλιώ υπάρχουν ρυθμίσει για όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν επικαλύψει. Δεν θέλω να γίνει τουλάχιστον αυτό με τη δική μου έκθεση. Και θα ήθελα τη βοήθειά σα και σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή. Εδώ αναφερόμαστε στο 70% του ΑΕΠ τη Ευρώπη και των ευρωπαϊκών θέσεων εργασία πάνω κάτω. Παρακαλώ λοιπόν, βοηθήστε μας να εστιάσουμε το πεδίο εφαρμογή, ούτω ώστε να έχουμε και προσταθέμενη αξία εδώ σε ό,τι αφορά την διέξοδο από την κρίση στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, άλλα κράτη-μέλη τα πήγαν καλά, άλλα υλοποίησαν σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχουν πολλέ φαιέ ζώνε όμω. Πρέπει να δούμε πώ λειτουργεί αυτή η αλληλεπίδραση με άλλε ε, νομοθετικέ πράξει. Και όλα βεβαίω εναπόκειται στι λεπτομέρειε, γιατί πρέπει να υπάρχει λόγο που η Επιτροπή έχει ε, κινήσει 12 διαδικασίε επί παραβάση. Πρέπει να βρούμε άλλου τρόπου μέσω του διαλόγου για να κατανοήσουν τα κράτη-μέλη ότι έχουν όφελο από την υλοποίηση, ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να είναι κάτι θετικό. Σα καλώ λοιπόν να μα βοηθήσετε να βρούμε και καλά παραδείγματα όπου η πλήρης ε, και σωστή και χρηστή υλοποίηση ε, και επιβολή της ε, οδηγίας περιπηρεσιών έχει επιφέρει προσταθεμένη αξία, έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Με θετικά και αρνητικά στοιχεία πάντα. Η Επιτροπή είναι σαφής ότι είναι βεβαίως μια εξαιρετικά καλή ανακοίνωση. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία με τον Επίτροπο Μπαρνιέ και πραγματικά εκτιμώ το γεγονός ότι πήγε, ταξίδευσε σε όλα τα κράτη-μέλη, ήρθε σε επαφή με του φορεί της αγοράς είδε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε αυτά τα νέα σημεία επαφή. Και εδώ θέλω να ακούσω και τις δικές σας απόψεις πώς μπορεί αυτό να γίνει διασυνοριακά. Η Επιτροπή, όπως είπα, ήταν σαφής. ...2,6% μέσα στα επόμενα 5-10 χρόνια είναι το εκτιμόμενο ε, ποσοστό. Και πραγματικά είναι μεγάλη η ευθύνη που μας αναλογεί. Περιμένω λοιπόν να ακούσω τις απόψεις σας και να λάβω κι εγώ ε, περισσότερες πληροφορίες ε, για την έκθεσή μου. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Να πω βεβαίως ότι ε, η κυρία Παριτέ ήταν η συγγύτρια για την αρχική έκθεση για αυτή την οδηγία και εγώ συνεργάστηκα μαζί της και βεβαίως και ξέρει πολλά σε αυτόν τον τομέα. Ας προχωρήσουμε τώρα στην πρώτη, στο πρώτο θέμα. Έχουμε τέσσερις ομιλητές. Ο κύριος Πέλκμας από το Κέντρο Ευρωπαϊκών Πολιτικών Σπουδών, το ΣΕΠΣ, είναι γνωστός για την ανάλυση όλων των πτυχών της ενισέας αγοράς και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες και ήταν ένας από τους πρώτους που με κάλεσε να επισκεφτώ τους φοιτητέ του όταν εγώ πρώτο ήρθα εδώ το 1999 ως πράσινος ευρωβουλευτής εδώ στις Βρυξέλλες. Τότε γνωριστήκαμε. Ήθελα λοιπόν να ακούσω τις απόψεις σήμερα. Ε, Έπειτα δώσουμε το λόγο στον Μέχτελ Ουμέν, αντιπρόεδρο της Business Europe και αναπληρωτή τη διευθυντή της Ομοσπονδίας ε, των Κάτω Χωρών ε, της επιχειρήσης. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτή την παρουσία και έπειτα έχουμε τον Τόμας Μάρεϊ που εκπροσωπεί την ε, Προεδρία του Συμβουλίου, Διευθυντή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Εξωτερικής Αγοράς, στο Υπουργείο Εργασίας, Επιχειρήσεων και Καινοτομίας. Χαιρόμεθα ιδιαίτερα για την παρουσία σας. Ε, και Ξέρουμε βεβαίω ότι η Πάτη Προεδρία έχει κάποιες ε, θέσεις σε κάθε αίθουσά μα ε, προ τα πίσω, αλλά σήμερα ειδικά η θέση είναι πιο κοντά στο Προεδρείο καθώς θα πάρει Και τέλος η κυρία Βερόνικα Νίλσον, γραμματέα της Ομοσπονδίας Συνδικάτων. σας υπενθυμίσω το ρολόι όταν αρχίσετε να το χρόνο, κάτι θα καταλάβετε, θα παρατηρήσετε το ρολόι να έρχεται πιο κοντά σας, τέλο πάντων ε, κάποια, κάποιο σημάδι. Και καλό είναι μετά την εισήγησή σα να ακούσουμε και κάποιε ερωτήσει από το κρατήριο και να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτέ τι ερωτήσει και να δώσουμε στο λόγο και κάποια καταληκτικά σχόλια. Ο κύριος Μπέλκμαν έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι πολλά τα 10 λεπτά για ένα περίπλοκο ζήτημα. Αλλά επειδή έχετε λάβει και διαφάνειες, θα σας καλέσω να τις παρακολουθήσουμε μαζί. Λοιπόν, σε τρία σημεία είναι χωρισμένη η εισήγησή μου, όπως είπε και η συγγήτρια. Κατά πόσον υπάρχει δυναμικό ανάπτυξης. Δεύτερον, η οικονομική έρευνα πώς μπορεί να μας εξυπηρετήσει καλύτερα στο άνοιγμα των Ινδοευρωπαϊκών αγορών υπηρεσιών. Έχω δύο διαφάνειες εδώ που μας, η πρώτη και η δεύτερη που θα δείτε, που εξηγούν κάποια πράγματα για την απασχόληση και εξηγούν πώς οι υπηρεσίες δεν είναι τομέας ανάπτυξης και δεν δίνει απασχολησιμότητα. Βλέπουμε λοιπόν ότι α, έχουμε αυτά τα στοιχεία. Βέβαια, οι υπηρεσίε έχουν έρθει αρκετά αργά στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, 55 χρόνια τώρα, βέβαια, για πολλού λόγου. Δεν έχουμε χρόνο τώρα να συζητήσουμε αυτό. Πάντω, το καλό των τελευταίων 10-15 ετών είναι ότι οι υπηρεσίε είναι κάτι που αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ σοβαρά μπαίνοντα και στο εθνικό επίπεδο. Δηλαδή, μια προσέγγιση σε δύο αν θέλετε, στρώματα ταυτόχρονα. Όμως πρέπει να ξεπεράσουμε τις υπηρεσίες για να καταλάβουμε και άλλα πράγματα, όπως θα πούμε και άλλοι α, ομιλητές. έτσι και λίγο καφές για να αυξηθεί και η παραγωγικότητά μου. Κατανοείτε, είναι και αυτή μια σημαντική υπηρεσία, λέει ο μιλητή. Λοιπόν, βλέπετε αυτή τη διαφάνεια γιατί είναι μια ε, περίληψη όλων όσων συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες. Αν θέλετε ένας πολύ σύντομος οδηγός, όπου βλέπετε το σύνολο των καθηκόντων στην πολιτική εναρμόνιση σε θέματα ανταγωνισμού κτλ. Βλέπετε την οδηγία των υπηρεσιών αριστερά πάνω και τέσσερα ρυθμιστικά καθεστώτα εκτός τις ε, οδηγίες των υπηρεσιών. Άρα είναι λάθος να εστιάζουμε μόνο στην οδηγία της υπηρεσίας. Να σας επισημάνω όμως ότι οι άλλοι τομείς, αν και ο τομέας μεταφορών είναι αρκετά μακριά, οι άλλοι τομείς, ρυθμιστικά καθεστώτα, πραγματικά ε, σημαίνουν ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο και με χαρά να σας ανακοινώσω ότι στην Ότχα Ευρώπη εγώ και ο συναδελφός θα παρουσιάσουμε ένα έγγραφο με τίτλο Enjoy the Single Markets for Network Industries στη Γαλλία. Ξέρετε, πριν από 20 χρόνια θα ήταν αδιανόητο, όμω τώρα αυτό μπορεί να γίνει για να δείτε ακριβώ πώ πρακτικά έχουμε επιτύχει τόσα αποτελέσματα αυτό το διάστημα. Με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Είναι επέπονο έργο, αλλά δίνει αποτελέσματα. Εδώ σε τη διαφάνεια βλέπετε την διαφορά ανάμεσα στο διασυνοριακό εμπόριο και υπηρεσίε και τι επενδύσει. Και εμπειρικά βλέπετε ότι έχουν να κάνουν μια μεγάλη διαφορά. Δυστυχώ το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο από το 2004 έως το 2006 πέρασαν ατέρμονες ώρες συζητήσεων, θα θυμάστε Πρόεδρε, ο πλευρά εμπορίου, ότι μακροπρόθεσμα το πιο σημαντικό θα είναι οι ξένε άμεσε επενδύσει. Αυτό σίγουρα θα είναι και όσο περισσότερο μακροπρόθεσμα. Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί και πρέπει να είναι ιδιαίτερα παρεμβατική για τις εγχώριες υπηρεσίες. Για πολλού λόγου, βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια, ακόμα και την Ονομισματική Ένωση, χωρί όμω να είναι αναγκαίο. Το ερώτημα που τίθεται είναι. Η οδηγία τη υπηρεσία ακριβώ αυτό κάνει η ε, σχολή και διεισδύει βαθύτατα στις εθνικές υπηρεσίες. Είναι πολύ μικρό το κομμάτι που παραμένει σε ευρωπαϊκό καθαρό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι πρέπει να τλούμε μαθηματικά διδάγματα όπως αυτή τη δεκαετία που βλέπετε να υποδεικνύεται στην ε, διαφάνεια 9 και πώς, με βάση τη βιβλιογραφία μπορούμε να δούμε πώς στο Miss ICT έχουμε πολύ μικρότερη πρόοδο από ό,τι από τις είπα το τελευταίο διάστημα. Κάτι που πρέπει να ξεχνάμε. Η μεταρρύθμιση των υπηρεσιών είναι πολύ σημαντική για τη βιομηχανία. Η σύνδεση είναι σημαντική. Θα δείτε και στην προηγούμενη διαφάνεια. Κοιτάξτε τις μπλε Η σημασία των υπηρεσιών στο μεταπληκτικό τομέα αυξάνουν σημαντικά και από πίσω υπάρχει και το πρόγραμμα πλαίσιο 7 και εκεί δείχνει, μπορείτε να δείτε πιο πολλές λεπτομέρειες ακριβώς για αυτή την πρόοδο. Έπειτα, σε χώριο εθνικό επίπεδο, την αυστηρότητα των κανόνων και τα PMR είναι τεχνικές μέτρησης ε, τον, να περθούν την περιοριστικότητα, αν θέλετε, και την αυστηρότητα αυτών των κανόνων. Τα PMR είναι δείκτες λοιπόν μέτρησης και μας δείχνουν ότι χαμηλότερα PMR, δηλαδή λιγότερο λιγότερα αυστηροί κανόνες, μακροπρόθεσμα δίνουν υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό μπορεί να μην το έχετε καταλάβετε άμεσα είναι πώς επηρεάζει άμεσα η υπηρεσία στη βιομηχανία. Το παράδειγμα που μπορώ να σας δώσω εδώ και θα καλύτερο είναι η Σουηδία που έχει τις λιγότερες συνέπειες από αυτό το, το φαινόμενο και η Αυστρία με, το, με τη μεγαλύτερη επιρροή. Καθώς αυτό το φαινόμενο είναι αρνητικό φαινόμενο καθώς επηρεάζει αρνητικά α, τη βιομηχανία με μεγάλο κόστος, ε, χρονοβόρες διαδικασίες, ε, παροχής υπηρεσιών κτλ. Και όλα αυτά ακριβώς σε μια χώρα που έχει πιο χρονοβόρες και ε, αργές υπηρεσίες. Βλέπουμε τις συνέπειες και στη μηχανία. Αν δούμε τώρα κάποιες μελέτες προσωμείωσης και βλέπετε παραδείγματα ε, παραγωγικότητας και πώς αυξάνουμε σε μια δεκαετία. Πώς σοβαρά βλέπετε τις μελέτες προσωμείωσης. Η προσωμείωση είναι πάντα μια προσωμείωση, αλλά στον δίνει αίσθηση αν υπάρχει πρόβλημα και πώς μπορεί να λυθεί. Και αν δούμε τις διαφορές στην αυστηρότητα αυτών των κανόνων από χώρα σε χώρα, μαζί μου κάποια εικόνα. Κάποια πράγματα μπορούν να επιληθούν μόνο σε εθνικό επίπεδο, κάποια άλλα προβλήματα μπορούν να επιληθούν μόνο από την οδηγία της υπηρεσία. Ένα άλλο ζήτημα, που ίσως αυτή την ακραίωση δεν είναι απόλυτα σχετικό, είναι η ρυθμιστική ετερογένεια. Αυτό δεν σημαίνει εγγενής ποικιλομορφία ή ότι τα κράτη-μέλη ρυθμίζουν το ίδιο πράγμα με το δικό τους καθαρά τρόπο δημιουργώντας τεράστια τερογένεια, χωρίς λόγο να υπάρχει αυτή η αναγκαστικά. Ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της τερογένειας, ή μάλλον αν, αν καταφέρουμε να εξαλείψουμε την ετερογένεια, οι συνέπειες θα ήταν εξαιρετικές και τεράστιες. για την Επιτροπή Ιστορική Αγορά είναι κάτι πολύ σημαντικό και να συζητηθεί αυτό και θέλω να καταγραφεί. Λοιπόν, Επτά συνέργειες οικονομικού χαρακτήρα έχει η οδηγία για τι υπηρεσίες. Επιτρέψτε μου ένα λεπτό. Συστήνω στην Επιτροπή σας και σε όσους ενδιαφέρονται να δείτε τις διαφάνειες 15 και 16 για να δείτε προσεκτικά όλες αυτές οι οικονομικές συνέπειες. Η έρευνα για τα σημεία 3, 4 και 5, ιδίω για τα 4 και 5, είναι σχεδόν μηδαμινή. Παρά τα αυτά, οι συνέπειε είναι σημαντικέ. Όπω βλέπουμε στι αλλοδαπέ θηγατρικέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντικέ συνέπειε, αλλά δεν έχουμε τα στοιχεία. Ξέρουμε ότι πολλέ είναι πιο αποτελεσματικέ από όλε τι κατηγορίε επιχειρήσεων. Μπορώ να προχωρήσω να δασκάλτικα στοιχεία. Ότι χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία από την έρευνα. Έπειτα υπάρχει η βιβλιογραφία για την αύξηση του ΑΕΠ και όταν υπήρχαν οι διαπραγματεύσεις για την οδηγία πριν από κάποια χρόνια, αυτές οι μελέτες ήταν ακόμη α, Και αυτή τη στιγμή έχουμε και την μελέτη της τα ΕΚΦΙΝ που αφορά την άρση των εμποδίων μόνο και μόνο από την οδηγία με μια άσκηση αμοιβαίας αξιολόγησης, βλέπετε στη δεύτερη κουκίδα. Και εδώ βλέπετε σε γράφημα τις ε, συνέπεις που θα έχουμε διασυνοριακά και σε επίπεδο ξένων άμεσων επενδύσεων. Και εδώ βλέπετε κάποιες λεπτομέρειες. Δείτε από όλα τα εμπόδια που υπάρχουν τι περιμένουμε να αλλάξει στο 2020 μέσα σε μια δεκαετία. Πράγματι η οδηγία περιμένουμε να μας δώσει πολύ προσδόρους καρπούς ακόμη. Τα συμπεράσματά μου είναι τα εξή. Οι μεταρρυθμίσεις των μέτρων υπηρεσιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο συνδέονται οικονομικά άρεκτα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υιοθετήθηκε η οδηγία, τα κράτη-μέλη προσπάθησαν να δείξουν συνεργασία, να κάνουν το screen, να κάνουν μια αξιολόγηση. Δεύτερον, α, αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα και την μηχανή και μόνο για τι υπηρεσίε. Τρίτον, για το ICT, κυρίω για τι βιομηχανίε χρήστε χρήστες του ICT είναι πολύ σημαντικό και τη σχέση μα με τη ΣΥΠΑ. Τέταρτον, χρειάζεται, υπάρχει άλλο μεγάλο περιθώριο ακόμα βελτίωση παραγωγικότητας, αν βελτιώσουν τα κράτη-μέλη το καθεστώς αυστηρότητας, χωρίς να απαλλαγούμε βεβαίως από ρυθμίσεις εντελώς. Και έπειτα να πούμε ότι υπάρχουν και Τομεί όπου υπηρεσίες δεν βελτιώνονται μόνο μέσω ανταγωνισμού. Χρειάζονται βαθιές επενδύσεις σε όλους τους τομείς και ιδίως υποδομέ. υποδομές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρος που καταφέρατε και ξεπεράσατε και τις προσδοκίες μου με το να μας προσφέρετε τόσο πολλά οικονομικά δεδομένα σε τόσο λίγο ε, χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι μας ζωγραφίσατε ένα ενδιαφέροντα πίνακα που θα μας βοηθήσει και θα αποτελέσει και το πλαίσιο για την υπόλοιπη ακρόαση. Θα παρακαλέσω την κυρία Όμεν τώρα. Των διαφανειών υπάρχουν αντίγραφα που θα πρέπει να τα έχετε κανονικά γιατί νομίζω ότι βέβαια έχουν μεγαλώσει οι οθόνες ε, τελευταία αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούν να είναι σχετικά μικρές για όσους θέλουν να τις παρακολουθήσουν μακρόθεν. Κυρία Όμεν, παρακαλώ. Πρώτα, ευχαριστώ την Επιτροπή σας και ιδίω την κυρία Μπίλτ που προσεκάλεσε το Business Europe να δώσει τις απόψεις της από την άποψη των επιχειρήσεων. Γνωρίζετε ότι εκπροσωπούμε μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και κάπως μεγαλύτερων, και θα ήθελα σήμερα να μιλήσω για τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι εταιρείε μας στην καθημερινή τους δραστηριότητα. Πρώτα που έχουν σχέση με την οδηγία υπηρεσιών, αλλά και πέραν αυτής. Θα αρχίσω λέγοντας ότι η οδηγία υπηρεσιών έφερε πολλά θετικά. Εξυγχρονισμό των δικαιωτικών πλαισίων, κατάργηση αδικαιολόγητων απαιτήσεων και αυτά είναι καλά. Ωστόσο, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν φραγμοί που αντιμετωπίζουν οι εταιρείε μας στην δουλειά που κάνουν και διαμεθοριακά. Και αυτό είναι κρίμα. Ο προλαλής αλλά και άλλοι είπαν προηγουμένως ότι υπάρχει ακόμα μεγάλο δυναμικό για ανάπτυξη και δεν μιλώ μόνο για τις υπηρεσίες, αλλά και για την βιομηχανία την ίδια. Γιατί υπάρχει και διασύνδεση, όπως εξήγησε και ο προηγούμενος ομιλητής, μεταξύ των δύο αυτών. το, δυναμικό λοιπόν οικονομικής ανάπτυξης είναι μεγάλο. Θα έρθω τώρα στους φραγμούς αυτούς που έχουν σχέση με την οδηγία υπηρεσιών. Αυτή είναι τριών ειδών. Πρώτα, υπάρχουν εμπόδια για τις επιχειρήσεις που θα έπρεπε να έχουν καταργηθεί ήδη από την ίδια την οδηγία υπηρεσιών. Και εδώ υποστηρίζουμε ακριβώς αυτή την πολιτική μηδενικής ανοχής. Δηλαδή να πάμε τις χώρες στα δικαστήρια. Στο δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άλλο είδος φραγμών έχει σχέση με την ελευθερία των χωρών μελών που τους έχει δώσει η Οδηγία Υπηρεσιών να διατηρήσουν ορισμένους περιορισμούς εφόσον τους θεωρούν αναλογικούς και δικαιολογημένους για λόγους ε, γενικού συμφέροντος. Εδώ ανοίγεται μια φαία ζώνη, μια γκρίζα ζώνη της οδηγίας υπηρεσιών. Ακούμε από επιχειρήσεις ότι καμιά φορά έχουν ερωτηματικά σχετικά με το εάν οι συγκεκριμένοι περιορισμοί θα πρέπει να διατηρηθούν για λόγους όντως δημοσίου συμφέροντος. Γιατί καμιά φορά πρόκειται απλώς για προστατευτικά μέτρα των τοπικών αγορών. Εμείς θεωρούμε ότι θα ήταν καλό να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια για το πώς χρησιμοποιούν την ελευθερία που τους δίνεται οι χώρες μέλη, διατήρησης δηλαδή περιορισμών για λόγους γενικού συμφέροντος και η λεγόμενη peer review που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ χωρών μελών δηλαδή και κομισιών εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα θετικό πρώτο βήμα. Όμως θα είναι καλό αυτό να γίνει πιο διαφανές. Δηλαδή πώς χρησιμοποιούν την ελευθερία αυτή που τους δίνεται οι χώρες Το 2009 και 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε ενημερωτικά σημειώματα στο Συμβούλιο για την πρόοδο της εφαρμογής της οδηγίας υπηρεσιών. Γιατί άραγε αυτό δεν γίνεται πλέον. Εμείς θεωρούμε ότι ήταν καλή ιδέα και θα πρέπει να ξαναγίνουν εκθέσεις από την Κομισιόν για το λεγόμενο State of Play προς το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, αλλά να διαβαστούν και στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά και να μπει και μία παράγραφος στα εθνικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το τρίτο είδος φραγμών που έχουν σχέση με την οδηγία υπηρεσιών έχει σχέση με τα points of single contact που εμείς θεωρούμε ότι προσφέρουν πλεονεκτήματα και στις επιχειρήσεις αλλά και στις κυβερνήσεις. Στις επιχειρήσεις διότι τους προσφέρουν πρόσβαση σε πληροφορίες αλλά και για να κάνουν τα γραφειοκρατικά επιγραμμικά online, αλλά και για τις κυβερνήσεις είναι σημαντικό γιατί έτσι εξυγχρονίζουν τις, δικη, τις δημοσίες δικήσεις τους, οδηγούνται και σε μείωση του κόστους χρησιμοποιώντας εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, e-government. Και αυτό επομένω εξοικονομεί χρήματα και για τις επιχειρήσεις και για τις κυβερνήσεις. Και εδώ ε, χωρεί βελτίωση. Και εδώ σημειώνω τρία πράγματα. Πρώτο, ότι η πρόσβαση σε καλές πληροφορίες μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη. Οι πληροφορίες αυτές να διατίθεται σε πλείονες γλώσσες, όχι μόνο της συγκεκριμένη χώρας μέλους, και τέλος, ότι οι εταιρείε, οι επιχειρήσεις να μπορούν να κάνουν όλη τη γραφειοκρατία επιγραμμικά. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα ότι η ελληνική υπογραφή, η signature, μα θα ήταν θαυμάσια να μπορούσε να λειτουργήσει σωστά και να χρησιμοποιείται. Έτσι λοιπόν σε εσά απευθύνουμε έκκληση να συνυπογράψετε έναν φιλόδοξο χάρτη πίεση και γιατί. Διότι θέλουμε να βελτιωθούν, να βελτιωθεί η λειτουργία των PSC και να δοθούν των points of single contact δηλαδή και επομένως να εξυπηρετηθούν καλύτερα επιχειρήσεις αλλά και οι κυβερνήσει. Τώρα ε, για τους φραγμούς που έχουν σχέση με την οδηγία υπηρεσιών αυτά ήταν. Τώρα το κύριο μήνυμά μου σήμερα είναι ότι εμείς πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όχι μόνο στόχευση στην ίδια την οδηγία υπηρεσιών αλλά και πέρα από αυτήν. Τι εννοώ. Εννοώ ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα και με άλλες οδηγίες και πρωτοβουλίες για παράδειγμα του ηλεκτρονικού εμπορίου ή των επαγγελματικών προσόντων αλλά και να εξεταστούν και άλλοι τομεί που δεν καλύπτονται ακόμη, ή δεν καλύπτονται μάλλον από την οδηγία υπηρεσιών, όπως ε, για παράδειγμα γραφεία προσωρινής έβρεσης εργασίας, ε, ασφάλειας. Να υπάρξει λοιπόν μια συγκεντρωτική, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Είπα λοιπόν ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ας γίνει και μια ανάλυση των υπολοιπωμένων φραγμών και να σας πω λίγα παραδείγματα από αυτά που αντιμετωπίζουν οι, υπηρεσί, επιχειρήσεις. Πρώτο παράδειγμα, αντιμετωπίζουν μεγάλο αριθμό προστατευμένων επαγγελμάτων, πάνω από 500, 800 μάλλον και 25 από αυτά σε μία μόνο χώρα μέλος. Για παράδειγμα, ο φωτογράφος γάμου ή ο μπάρμαν είναι ρυθμισμένο επάγγελμα. Αυτό μας προκαλεί κάποια ερωτηματικά. Είναι για απαραίτητο. Ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φτιάξει ένα κατάλογο των ρυθμισμένων επαγγελμάτων. Και οι χώρες μέλη ας αναλάβουν κάποια δράση για να μειωθούν αυτά τα ρυθμισμένα επαγγέλματα που στο κάτω της γραφής είναι όντως εμπόδιο για την άσκηση δραστηριότητα των επιχειρήσεων και επίσης υπάρχει και εξακολουθεί και υπάρχει έλλειψη αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Δεύτερο παράδειγμα, θέματα διπλής ασφάλειας. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση πρέπει να είναι ασφαλισμένη σε μία χώρα μέλος, αλλά μετά τη ζητούν να ασφαλιστεί και σε άλλη χώρα μέλος. Αυτό κοστίζει και χρόνο και χρήμα. Τρίτο παράδειγμα φραγμού είναι ότι υπάρχουν πολλά αντικρουόμενα εθνικά πρότυπα και έλλειψη αμοιβαία αναγνώρισης στον τομέα των αγαθών. Είναι πολύ σύνηθες να υπάρχει αυτή η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, όχι όμως στις υπηρεσίες. Εμείς θεωρούμε ότι θα είναι καλύτερο γιατί θα αναπτυχθεί και εμπιστοσύνη και κατανόηση με την αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των χωρών μελών. Για παράδειγμα, για την διαπίστευση ειδικών και για την κύρωση πιστοποιητικών. Άλλο που αναφέρθηκε και πριν για τη χωροταξία. Ακούμε από τις επιχειρήσεις μας ότι καμιά φορά εμποδίζονται από αυτό που ε, ονομάζουμε στα αγγλικά economic, needs test. Και ένα πέμπτο απαιτήσει νομικές και κυριότητας όταν ε, δηλαδή θέλουν να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα μέλος και τέλος έλλειψη παραγωγικότητας σε επιχειρηματικές υπηρεσίες όπως για παράδειγμα πληροφορικής και επικοινωνιών, ε, προσφράση υπηρεσιών σε άλλες επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει καμιά ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στους τομείς αυτούς. Και θα είναι καλό ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή εν πάση περιπτώσει εμείς υποστηρίζουμε την ίδρυση ενός, μιας μάλλον ε, ε, ομάδας υψηλού επίπεδου για τις υπηρεσίες business to business και να δουν τι ακριβώς απαιτείται εκεί. Αυτά λοιπόν με λίγα λόγια ως επισκόπηση ορισμένων από τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι ε, επιχειρήσεις στην καθημερινή ζωή και ελπίζουμε ότι θα κατανοήσετε ότι πραγματικά πρέπει τώρα πια να αναλυφθεί δράση και να γίνουν βήματα για να ολοκληρωθεί η αγορά των υπηρεσιών στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζουμε ότι πρέπει να ληφθούν τρία βήματα, να, τρία μέτρα, να γίνουν τρία βήματα. Να επιβληθεί η υπηρεσία, ε, συγγνώμη, η οδηγία υπηρεσιών, μηδενική ανοχή στους φραγμούς και ανάλυση των φραγμών για το πώς θα αντιμετωπιστούν και τρίτο, αμοιβαία αναγνώριση και αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των χωρών μελών. Εμείς απευθύνουμε έκκληση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει πίεση με τη σειρά του στις χώρες μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία υπηρεσιών. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας προσφέρατε να σας αναπτύξουμε ε, το θέμα εκ μέρους των επιχειρήσεων. Βεβαίως μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα. Αλλά πάντως εμείς συντάσσουμε έκθεση με συγκεκριμένα στοιχεία για τα εμπόδια αυτά και θα σας την διαβιβάσουμε. Ευχαριστώ. Well, thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι πολύ επίοικη σήμερα το απόγευμα, Συνήθω αυτό δεν ισχύει, αλλά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσε οι παρουσιάσει σας. Τώρα, καλά τα μας στο βήμα για να μας κάνετε δική του παρουσίαση σε ό,τι αφορά την οδηγία υπερυπηρεσιών. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Αννα Μαρία που ε, έθιξε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Με τα και προσωπώ την ε, Προεδρία και καθώς προέρχομαι και από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, Μπορώ να σα πω ότι είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση χθε ε, στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα. πολιτική συζήτηση ε, για την ολοκλήρωση τη ενιαία αγορά ε, και για την υπηρεσία, για την οδηγία περί και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την υλοποίησή της στα κράτη-μέλη. Και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της αιτήσεις έκθεσης πρόοδου. Κάτι στο οποίο συμφωνήσαμε όλοι και μπορούμε να εξετάσουμε και πολλές μελέτες που έχουν εκπονηθεί αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις της οδηγίας υπηρεσιών. Δηλαδή ότι ε, η εφαρμογή της οδηγίας θα βελτιώσει το ε, περιβάλλον για τους παρόχους υπηρεσιών μέσω της μείωσης του διοικητικού άχθους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας και του εύρους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και ως εκ τούτου και με μείωση των τιμών. Αυτό είναι δεδομένο. Οι μελέτες, οι πρόσφατες μελέτες ε, από το Ολλανδικό Γραφείο Εμπορικής Πολιτικής, Οικονομικής Πολιτικής έχει δείξει ότι ε, οι υπηρεσίες αυτές θα μπορούσαν να τριπλασιαστούν αν εξαφανίζονταν εντελώς οι διαφορές ε, στην εφαρμογή. Οι εξαγωγείς μας βεβαίως συνδέονται και με την εσωτερική αγορά και με την παγκόσμια αξιακή αλυσίδα. γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστια σημασία σε ό,τι αφορά το διεθνέ εμπόριο και τι επενδύσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο μεγαλύτερο εξαγωγέα, εισαγωγέα, πηγή και παραλήπτη ε, των ε, έμεσων ξένων επενδύσεων. Αν όπω περιμένουμε το 90% τη οικονομική δραστηριότητα μέχρι το 2015 ε, παρουσιαστεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς όλοι έχουμε, θεωρούμε απαραίτητο να μείνουμε στο ίδιο μήκο κύματο προ όφελο των καταναλωτών μα. Πρέπει βεβαίω να οικοδομηθεί μια ενιαία αγορά ω ε, ένα φορέα ενοποίηση και δεν έχουμε κατακτήσει ακόμα αυτό το βέλτιστο επίπεδο. Και γι' αυτό και η οδηγία περί έχει ενσωματωθεί σε ολόκληρη την εμπορική ε, ατζέντα, το εμπορικό θεματολόγιο. Και λόγω της ε, οικονομικής κρίσης και στην Ευρωζώνη το όλο πρόγραμμα που αφορά την ενιαία αγορά ε, περνά μια πολύ δύσκολη θέση, φάση, υπάρχει κίνδυνος ε, στασιμότητας και οπισθοχώρησης. Γι' αυτό και απαιτείται μια στενότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Για τα στατικά στοιχεία περί πράγματι ήταν ε, αξιοθαύμαστα αυτά τα στατικά στοιχεία αναφέρθηκε το ποσοστό 70-71% του συνολικού ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3,2% μόλις αυτού ε, προκύπτει από την ενδοευρωπαϊκή εμπορική δραστηριότητα. Και αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, γιατί ε, οι εμπορικέ σχέσει ισοδυναμούν με την ανάπτυξη και τι θέσει εργασία. Βεβαίω, απαιτείται τεράστια πολιτική βούληση και δέσμευση και να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσει. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις οικονομικές αυτές ε, ανάγκες, τη γραφειοκρατία, το, την απελευθέρωση επαγγελμάτων, διοικητικές απαιτήσει για ε, ξένους παρόχους. Οι δυσκολίες βεβαίως είναι σημαντικές. Ο αντίκτυπος στο ΑΕΠ θα μπορούσε και πάλι να ποικίλει μεταξύ 0,6% και 1,5% ή για να το πω πιο συνολικά, μέχρι και με 400 δις ευρώ θα μπορούσαν να φτάσουν οι επιπτώσεις. Αναφέρθηκε το 7 και 4% προηγουμένως. Τα ωφέλη τώρα από την ε, περαιτέρω απλούστευση και την άρση των φραγμών είναι εξίσου σημαντικά. Αδιαφεσβήτητα υπάρχουν κάποιες ε, υποχρεώσεις που προκύπτουν από την υπηρεσία και φτάνουν όλα τα επίπεδα ε, διοίκησης, κυβερνητικής διοίκησης. Δεν είναι μόνο σε εθνικό ή ευρωπαϊκό ε, θέμα, φτάνει ακόμα και στο τοπικό επίπεδο, υπερφυριακό. Ωστόσο, αυτή η συστηματική αλλά και συστημική υλοποίηση του συνόλου των κανόνων που προκύπτουν από την υπηρεσία από την Οδηγία Περιπηρεσιών αποτελεί τεράστια πρόκληση για τις αρχές των κρατών μελών, ιδίως για τα κράτη-μέλη που έχουν ένα πιο αποκεντροποιημένο σύστημα διακυβέρνησης και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα τελευταίε δύο ημέρε ε, συζητεί την ετήσια έκθεση προόδου και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Για πρώτη φορά, η ολοκλήρωση τη ενιαία αγορά και η υλοποίηση τη οδηγία υπηρεσιών ε, αποτελούσε τμήμα αυτής της συζήτησης και αυτό είναι πολύ καλό σημείο κίνησης και με τα χαράς μπορώ να πω ότι όλα τα κρατημέλη δέχθηκαν και χαιρέτησαν την ε, ενσωμάτωση αυτού του τομέα πολιτικής ε, στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και όλα τα κρατημέλη τουλάχιστον αυτά που πήραν το λόγο, η πλειονότητά τους δηλαδή, επικρότησαν και την ενσωμάτωση της, ενσωμάτωσης, της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς στην όλη διαδικασία. Αυτό τώρα θα περάσει στις συστάσεις, στις ειδικές αναχώρα συστάσεις και θα αποτελέσουν τμήμα των ε, υποχρεώσεων των κρατών μελών για να ολοποιήσουν και τις ε, διατάξεις ε, της οδηγίας περιπηρεσιών. βασίστηκε και σε ένα έγγραφο που προέκυψα από προηγούμενη συνεδρίαση υψηλού επίπεδου η οποία τόνισε ότι πάλι πρέπει να υπάρξει η συνέχιση ε, της ε, συστημικής και συστηματικής ε, υλοποίησης της οδηγίας, αλλά και για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και η χρήση της αξιολόγησης ομοτήμων, του peer review, ελήφθη υπόψη. Πολλοί από τους φραγμούς δεν είναι φυσικοί πραγματική δηλαδή, αλλά περισσότερο διοικητική. Και είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν ξεκάθαρα. Και έτσι κάποια κράτη-μέλη για, σε ό,τι αφορά ας πούμε το, την ενιαία θηρίδα ε, τα έχουν υλοποιήσει καλύτερα, Κάποιοι τα έχουν υλοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό, κάποιοι σε μικρότερο λοιπόν. Όπως αν θέλετε, υπάρχουν ε, κάποιοι πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα. Σε περιπτώσεις όπου έχει αναπτυχθεί τέτοιο σύστημα, υπάρχει πληθώρα ε, κυβερνητικών ε, ιστοτόπων και, και πυλών. Και αυτό βοηθάει και στην υλοποίηση της ε, οδηγίας. Σε αντίθεση με αυτό, άλλα κράτη-μέλη είχαν σημαντικά προβλήματα να επιλύσουν ό,τι αφορά την ανάπτυξη των ε, single points of contact και των ηλεκτρονικών ε, συναλλαγών. και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της πολιτικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Και αυτό έχει πολύ επιπτώσεις. Κάτι το οποίο επιφέρει και περαιτέρω δαπάνες, βεβαίω που δεν είναι ευχάριστο σε τέτοιε περιόδους. Απαιτείται περαιτέρω, απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την ε, άρση αδικαιολόγητων ε, εμποδίων φραγμών, ιδίω ό,τι φορά το λιανικό εμπόριο, τα ε, περιορισμένα επαγγέλματα, τις κατασκευές και την βιομηχανία και τα peer reviews εκεί έδειξαν ότι υπάρχει ένας τέτοιος στόχος. Οι ειδικέ ανασυστάσεις σε χώρα θα αναφέρουν και την απελευθέρωση ορισμένων επαγγελμάτων, ότι δηλαδή κάποια κράτη-μέλη θα πρέπει να αναθεωρήσουν ή να αξιολογήσουν την εγχώρια νομοθεσία. Είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο. οι επιχειρήσει και πάλι έρχονται αντιμετώπιση με μεγάλο βαθμό γραφειοκρατία. Εξακολουθούν να ισχύουν οι εθνικοί κανόνε. Κάποιε φορές υπάρχουν και φραγμοί που συνδέονται με τον, ε, με τον έλεγχο τη οικονομική ανάγκη, κατά πόσο δηλαδή χρειάζονται περαιτέρω φορείς ή όχι. Τώρα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο υπάρχουν πραγματικά τέτοιοι φραγμοί ανακλάδο. Ίσως χρειαζόμαστε μια πιο επικαιροποιημένη οικονομική ανάλυση για αυτούς τους ε, κρίσιμους ε, τομείς και σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει και μια ειλικρίνη από πλευράς κατομελών και περαιτέρω διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Πολλές ε, συμβουλευτικές ομάδες υψηλού επίπεδου αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένους τομείς όπως ο χάλιβας, ε, τα αγροτικά προϊόντα και Η Επιτροπή πολύ γρήγορα σύστησε ε, μια αντίστοιχη ομάδα υψηλού επίπεδου για τις επιχειρήσεις και τι υπηρεσίε, με υψηλή συμμετοχή και σίγουρα και η Ιρλανδική Προεδρία το θεωρεί προτεραιότητα. Περιμένω λοιπόν με ανυπομονησία την ε, έκθεση της συγγήτριας και ελπίζω και εγώ να συνέβαλα σε ένα βαθμό. Ευχαριστώ. Να πατήσω στον εκπρόσωπο της Ιρλανδικής προεδρία κατά τη συζήτηση να προετοιμαστείτε να είστε πιο συγκεκριμένο. Σα το λέω από τώρα για να το σκεφτείτε. Right. We've got... We haven't started the questions yet. Δεν ξεκινήσαμε ακόμα τον κύκλο των ερωτήσεων, λέει ο Πρόεδρος. Ο κ. Μάρη πολύ ορθά μίλησε για κάποια εμπόδια Βλέπετε όμω, εγώ βλέπω κάποιο τίτλο εφημεριδών που λέει ότι στο Alba που ίσω να μην το γνωρίζετε, όπου έλαβαν χώρα χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνε, από ό,τι φαίνεται, ενημέρωσαν αθλητές τους και ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. 5.000 εργασίε θα χαθούν, λένε οι εφημερίδες αυτά θα τα περάσω στον κύριο Μπαρνέ για μια αμοιβαία συνεργασία τέτοιων θεμάτων. Κύριε Νίλσον, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι μαζί σας και θέλω να σας συγχαρώ επίσης για την σχεδόν εξαιρετική ισορροπία μεταξύ των δύο φίλων στην εκπροσώπησή τους. Εγώ θα ε, προσεγγίζω το θέμα από διαφορετική οπτική γωνία, αν θέλετε μια πιο κοινωνική οπτική γωνία. Θέλω να επενθυμίσω πρώτα απ' όλα ότι η ενιαία αγορά και τις υπηρεσίες δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι εργαλείο για την επίτευξη κοινωνική προόδου, για την ε, καλή διαβίωση των εργαζομένων, των πολιτών, των επιχειρήσεων. Κάτι πολύ σημαντικό που να ξεχνάμε όταν κάνουμε αξιολόγηση τη εφαρμογή τη οδηγίας για τις υπηρεσίες. Και καλούμε τα κράτη-μέλη να μελετήσουν σε μεγαλύτερο βάθος συμβολή τη ιστορικής αγορά σε αυτό το στόχο και να κάνει και η Κομισιόν μια αξιολόγηση αυτών των μέτρων ε, που έχουν εφαρμοστεί ως τώρα. Πάντα υπάρχουν καλά και κακά παραδείγματα. Όσο είναι υπέρ των θα βρουν καλά παραδείγματα. Όσο είναι κατά θα βρουν τα κακά παραδείγματα. Χρειάζεται λοιπόν μια κάπω αν θέλετε ουδέτερη αξιολόγηση των πεπραγμένων έω τώρα στον τομέα. Παρότι η εφαρμογή της οδηγίας ε, για τις οδηγίες οδήγησε στην άρση πολλών εμποδίων. Εμπόδια παραμένουν ακόμη και σήμερα. Ακούστηκαν από προλαλήσατες κάποια από τα εμπόδια αυτά, όμως το μέσο των υπηρεσιών πραγματικά είναι μεγάλος, περιπλοκός και σίγουρα πετύχει χρόνο για να εναρμονιστεί όλη η ευρωπαϊκή αγορά μέσω ευρωπαϊκή Νομοθεσία και η οδηγία αυτή δεν έχει εφαρμοστεί πλέον εδώ και τόσο πολύ καιρό. Συμφωνώ λοιπόν με τα συμπεράσματα της Κομισιόν να μην ξανανοίξουμε και πάλι ε, την οδηγία τουλάχιστον όχι τώρα. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι ε, το επίκεντρο της συζήτησης είναι πώς θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Θέλουμε μια νέα αγορά για τις υπηρεσίες να συμβάλλει θετικά στην αποσχολησιμότητα τα ποσοστά ανεργίας ε, είναι ρεκόρ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά τα ποσοστά για τους νέους είναι δραματικά υψηλά. Υπάρχει ένα κίνδυνος να χαθούν γενιές ολόκληρες λόγω αυτής της κρίσης. Και παρότι λέμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο τέλος της κρίσης, ακόμη δεν είμαι τόσο σίγουρη με τις προβλέψεις ε, της Κομισιόν ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μας λέει πως ναι, αλλά ε, υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμη αν δούμε ότι χρειάζεται πάντοτε πιο πολλούς χρόνους για να περάσει, αν θέλετε, κάποια ε, θετική αλλαγή και στην αγορά εργασίας. Και εκεί διαφωνώ με την εισηγήτρια. Δεν πιστεύω ότι μπορείς να διαχωρίσεις τη δημιουργία θέσεων εργασία με τι συνθήκε εργασία. Φοβούμαι ότι πολλέ από τι νέε θέσει εργασία που δημιουργούνται στο τομέα των υπηρεσιών είναι χαμηλών δεξιοτήτων, είναι μονότονε και πολύ κακά αμοιβόμενε. Βλέπουμε μία αύξηση του αριθμού των φτωχών εργαζομένων και είναι κάτι που σε καμία δεν βοηθά στη βελτίωση της ε, ζωής των εργαζομένων. Έπειτα, η ποιότητα της απασχόλησης είναι σημαντική και για έναν άλλο λόγο επίπεδα μισθών, συνθήκες εργασίας που επηρεάζουν και την ίδια την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται. Κακές συνθήκες εργασίας οδηγούν πολύ συχνά και σε κακές υπηρεσίες. Ε, σημείωσα και με ενδιαφέρουν επίσης την πρόταση της Κομισιόν για μία ανεκτική πολιτική για μηδενική ανεκτικότητα όταν δεν υπάρχει εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Πράγματι είναι σημαντικό αυτό. Δεν διαφωνώ μεν, αλλά η μηδενική ανεκτικότητα θα πρέπει να ισχύσει και σε άλλους τομείς. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τομείς όπου η Κομισιόν δεν ξεκινά διαδικασία επί παραβάση, αν και θα μπορούσε για την οδηγία τη υπηρεσία να το κάνει, αλλά ισχύει αντίστοιχα και για άλλους τομεί αυτό. Άλλοι τομεί, που έχω στο μυαλό μου, όπως η παραβίαση της αρχής της ελευθερίας εγκατάστασης. Πολύ συχνά αυτό χρησιμοποιείται και ως δικαιολογία για την πρόσληψη εργαζομένων και ειδικά φθηνού εργατικού δυναμικού η αρχή της χώρας ε, του εργαζομένου θα πρέπει να ισχύει για να εφαρμόσει, ε, μάλλον να μπορεί να προστατεύσει τους ε, εργαζομένους και τους καλή την πίστη εργοδότες ώστε να μην γίνεται παραβίαση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα εργατικά. Επειδή θα πρέπει να υπάρχει παραβίαση των κανόνων που ισχύουν αυτή τη στιγμή και μέσω της οδηγίας για τις υπηρεσίες και θα πρέπει να, υπάρχουν, να εφαρμοστούν μάλλον αποτελεσματικές κυρώσεις από την Κομισιόν για αυτές τις παραβιάσεις. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να μην είναι κατάλληλη ε, και αντίστοιχη η μισθή των εργαζομένων ή κάποιες φορές να ξεχνιόνται, αν θέλετε το πω έτσι, τροποντινά ε, να καταβάλλονται κοινωνικές εισφορές των εργαζομένων στόχος της οδηγίας είναι να αντιμετωπίσει τις ε, καταχρήσεις ε, και να, μεταξύ άλλων, θα λέγω ότι πολλά από αυτά που μπορεί να κάνει ε, η Επιτροπή μέσω της οδηγίας των υπηρεσιών μπορεί να τα κάνει ήδη και με άλλους τρόπους και σας καλώ και εσείς να βοηθήσετε ώστε αυτή η οδηγία να έχει νόημα για τους αποσπασμένους εργαζόμενους που τόσο πολύ ε, ευαγγελίζεται ότι θέλει να υπερασπιστεί. Δεν θα πρέπει λοιπόν να λειτουργεί διαφορετικά και αυτό ειδικά θέλω να πω ισχύει για το άρθρο 9. Θα πρέπει να υπάρχει ανοιχτός κατάλογος για τα εθνικά μέτρα ελέγχου, θα πρέπει να είναι δεσμευτικό κατάλογο, η κείμενη κατάσταση δεν θα βελτιωθεί τέλος. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ επίμαχο αυτό που θα πω και θα διαφωνήσετε πιο πολύ, αλλά θα επιμείνω. Θα επιμείνω στο θέμα της κοινή αστικής ευθύνης, γιατί μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε τις καταχρήσεις που βλέπουμε σήμερα και θέλουμε να το αποφύγουμε όλοι. Για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό. Επίσης θέλω να αναφερθώ στον κανονισμό Μόντι γιατί αυτό ήταν μια προσπάθεια της Κομισιόν να διευκρινίσει, να ξεκαθαρίσει ε, το ζήτημα της άσκησης του δικαιώματος ε, της ελεύθερης εγκατάστασης και της παροχής υπηρεσιών. το Μόντι 2 έχει αποσυρθεί. Υπάρχει η διαδικασία την κάρτα που ξεκίνησε από πολλά εθνικά κοινοβούλια. Οι κοινωνικοί εταίροι είναι δεσμευμένοι με την πρόταση και χαιρετίζουμε την απόσταση της πρότασης. Όμως τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τις αποφάσεις του Ευρωκοδικαστηρίου υπάρχουν γιατί οι αποφάσεις ισχύουν. Ότι η πρόταση της Κομισιόν δεν είναι ικανοποιητική δεν σημαίνει ότι σηκώνουμε τα χέρια και δεν κάνουμε τίποτα. Στην πρότασή μας, μάλλον η πρότασή μας είναι ένα πρωτόκολλο κοινωνικής πρόοδου που θα πρέπει να το επισυνάψουμε στις συνθήκες, ότι δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα υπερέχουν των οικονομικών ελευθεριών, αν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ αυτών. Ξέρω ότι τα θέματα όλα αυτά συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους και θέλω να πω και κάτι για την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα που ανέβηκε ο συναδέλφος από την Business που Χαιρετίζουμε την οδηγία αυτή, είναι πολύ σημαντική. Θα βοηθήσει τη δυσλογική κινητικότητα και πιστεύουμε ότι θα έρθουν κάποια από τα θέματα, τα εμπόδια που αναφέραμε και πριν. Τέλος, θα, εμείνω στα, θα τα, το κρατήσω τώρα των 10 λεπτών, αλλά θέλω να πω εν τέλει ότι είναι πολύ σημαντική η κοινωνική διάσταση της όλης της συζήτησης. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να παραγνωρίζουμε. Επίσης, η καλύτερη λειτουργία τη εσωτερική αγορά και τη υπηρεσία δεν είναι η μόνη λύση για την εντόμηση τη κρίση, γιατί συνεχώ μιλάμε για την κρίση. Για να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη και απασχολησιμότητα, θα πρέπει να σταματήσουν και πολιτικέ λιτότητε από τι κυβερνήσει. Δεν είμαστε κατά ε, τη οικονομική εξυγίανση, αλλά είναι πλέον καιρό ε, να αλλάξει αυτή η πολιτική. Ήδη ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μειώσουν το δημοσιονομικό του έλλειμμα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται μια μέρα στην άλλη. Και δεν μπορεί αυτό να γίνει στι πλάτε των εργαζομένων. Ανταπόκριση στην κρίση, είπαμε ναι, άρση των εμποδίων, αλλά όχι πάντοτε ε, στην πλάτη των εργαζομένων. Επενδύσει. Θέλουμε ευρωπαϊκά προγράμματα επενδύσεων και να σταματήσουν τα μέτρα λιτότητα. Αυτά είναι κάποια τα μέτρα που χρειάζονται για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση. Ευχαριστώ πολύ. thank you very much. Uh, Ευχαριστώ και τους τέσσερις. Ας ακούσουμε τώρα ερωτήσεις και σχόλια συναδέλφων. Πρώτα τους και οδησίγητες. Φαντάζομαι ότι οι σκιώδεις θα θέλουν να λάβουν επιστολόγο όπως η κυρία Ράπτη και εγώ θα δούμε τώρα ίσως να μην δώσω λόγο στον εαυτό μου, χρόνο στον εαυτό μου η κυρία Κοράτσα Μπίλτ παρενέβη πριν ας ακούσουμε πρώτα τους Αννα Αναμαρία και μετά έρχομαι Ας ακούσουμε πρώτα την κυρία Ράπτη λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ακούσουμε ε, την κυρία Γκέπχαρτ, την εξαίρετη συνάδελφο που έχει εργαστεί για αυτή την οδηγία και έχει πολύτιμη εμπειρία που νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει και δεύτερον διότι θεωρώ εξίσου σημαντική τη δική σας εμπειρία και συμβολή στην εργασία μας και άρα θέλω, θα ήθελα οπωσδήποτε να ακούσω και την δική σας κουβέντα. Λέω λοιπόν πάρα πολύ σύντομα ε, σε σχέση με την Business Europe. Ε, καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που είναι σήμερα εδώ και μας δίνουν το χρόνο τους καταρχήν και τις πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες τους. Επίσης, ε, να ευχαριστήσω την Άννα, Μαρίνα, Μαρία Κοράτσα Μπίλτ για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα, ε, για την δυναμικότητά της η οποία α, μας κρατάει πραγματικά σε γρήγορση και άρα να δουλέψουμε και να κάνουμε το καλύτερο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, θέλω επίσης να δώσω συγχαρητήρια στη Γραμματεία και τον Πρόεδρο της Επιτροπής για το εξαιρετικό hearing το οποίο διοργανώνεται, διότι μετέχουν όλες οι φωνές, όλες οι απόψεις. Ρωτώ λοιπόν, ε, την Business Europe, το ερώτημά μου είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Το άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω τόπου κατοικίας ή υπηκότητας του καταναλωτή. Ρωτώ, πώς πιστεύετε ότι μπορούν να υποστηριχθούν καλύτερα οι επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως είναι η ασφάλεια δικαίου και οι διαφορετικές γλώσσες στο διασυνοριακό εμπόριο. Θέλω να ρωτήσω την Προεδρία τι περιθώριο έχει στον περιορισμένο χρόνο της στην, στο πιδάλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει μία όθηση στην καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας διασφαλίζοντας την προστασία και των καταναλωτών και των εργαζομένων. Και τρίτο και τελευταίο θέλω να ρετήσω την εκπρόσωπο της ΕΤΟΚ ε, ποιο πιστεύει ότι θα είναι το αποτέλεσμα της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περαιτέρω απελευθέρωση και χαλάρωση του κανονιστικού πλαισίου. Ευχαριστώ. Σημαντικά ερωτήματα, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλοί ομιλητέ, πολλές ερωτήσεις, έτσι θα είμαι σύντομο. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσει σα που ήταν συνοπτικές και σημαντικά στοιχεία. Μία διευκρινιστική ερώτηση προς την κυρία Όμεν. Για το θέμα της εφαρμογής. Λέτε ότι ακόμα δεν εφαρμόζεται πλήρως ούτε ορθά. Και αναφερθήκατε σε αποφάσεις. Επειδή χθε ακούσαμε για τα βαθμολόγια μας, τα scoreboard, σχετικά με το επίπεδο εφαρμογής και το νέο ρεκόρ είναι 0,6 που φαίνεται να είναι πολύ ωραίο και καλό νέο για την διαδικασία. Μπορείτε να πείτε πιο συγκεκριμένα πού έγκυται το πρόβλημα και πού βλέπετε εσείς να μην εφαρμόζετε, αφού φαίνεται να τα πηγαίνουμε καλά με την εφαρμογή. Εγώ ως και θα μιλήσω αργότερα. Α, ο κύριος Έντερ, συγγνώμη, ναι. Είστε τόσο πίσω από την ενωτική αριστερά. Σύντομη παρατήρηση. Δεν μπορώ να φανταστώ να συζητούμε βελτίωση της οδηγίας υπηρεσιών χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τους ανθρώπους τους ίδιους και τις ανάγκες τους για δουλειά. Τι γίνεται με την ποιότητα της εργασίας, με τη μεταχείριση των ανθρώπων και με την αμοιβή τους. Μου φαίνεται παράλογο ότι συζητούμε εδώ ανεξάρτητα από τις ανάγκες των ανθρώπων. Δεύτερο, το ζήτημα της κατάχρησης που τόνισε ιδιαίτερα η κυρία Νίλσεν. Παίζει ωστόσο σημαντικότερο ρόλο από όσο έχει συζητηθεί μέχρι τώρα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη Γερμανία έχουμε ολόκληρο αριθμό ε, συμβουλευτικών υπηρεσιών που έχουν να σας πούν πάρα πολλά για περιπτώσεις καταχρήσεων σε σχέση με την οδηγία υπηρεσιών με οδηγίες, με, συγγνώμη, με, με εταιρείες που έχουν μόνο ένα γραμματοκιβώτιο ως διεύθυνση και ούτω καθεξής. Και εδώ μιλώ για την προστασία των ανθρώπων. Εμένα μου έρχονται καταγγελίες από επιχειρήσεις για την οδηγία υπηρεσιών και την κατάχρησή της για αθέμητο ανταγωνισμό σε περιπτώσεις υποβολής διαγωνισμών ε, τοπικών ή κοινοτικών αρχών κλπ. Απάτες δηλαδή. Δεν είναι μόνο το θέμα αυτό. Είναι και ζήτημα ισότιμων όρων ανταγωνισμού για επιχειρήσεις στον τομέα Παροχή υπηρεσιών και για παράδειγμα στον τομέα της οικοδομής. Και αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη στη συζήτηση τη Παγκόσμιας επιτροπή. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος Χάρμπορ. Έχω και εγώ ορισμένε ερωτήσει για κάπω αργότερα. Αλλά θα ακούσω πρώτα άλλους βουλευτές. Και θα φροντίσω ώστε να απαντηθούν όλες οι... Θα σας πω τα ονόματα Είστε στη λίστα, μην ανησυχείτε. Λόγκεγκάρντ. Διαδικαστικό. Μήπως μπορείτε να κάνετε ομάδες τριών ερωτήσεων και μετά να απαντήσουν. Ναι, δεν θα προλάβω, έχω και άλλους δύο. Θα δούμε. Αν οι ερωτήσει που κάνετε είναι μακροσκελήσει, τότε... Όπερ Όπερμαϊρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ για τις ε, παρουσιάσεις. Αναφέρομαι κυρίως στην πρώτη και επειδή αναφέρεται και η πατρίδα μου η Αυστρία, έχει για μένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρώτο, φαίνεται ωραίο αυτό το knock-on effect και τα λοιπά, γιατί θα διευκολυνθεί ε, η ανάπτυξη της οικονομίας κτλ. Τίθεται το ερώτημα κατά πόσον διατηρούνται τα κοινωνικά, οι κοινωνικές προδιαγραφές που είναι και διαφορετικές μεταξύ των χωρών μελών και κατά πόσον έχουν ληφθεί υπόψη στην μελέτη που αναφέρατε. Εγώ νομίζω πως όχι. Δεύτερο, για το παράδειγμα της Αυστρίας που λέτε ότι υπάρχει χαμηλός ανταγωνισμός λόγω υψηλών φραγμών λόγω της αργής εφαρμογής της οδηγίας. Λέτε ότι μπαίνει εκεί το θέμα της δημόσιας διοίκησης. Εγώ νομίζω ότι εδώ υπάρχουν ή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλα. Η συνολική οικονομία. Αναφέρατε το παράδειγμα των καπνόδοχων καθαριστών. Θα σας πω ένα παράδειγμα που δεν έχει μόνο σχέση με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, ο καπνόδοχο καθαριστής δεν είναι, έχει μονάχα το καθήκον να καθαρίζει την καπνοδόχο, έχει και σημαντικό ρόλο στην πρόληψη πυρκαγιών. Είναι και πραγματογνώμων. Επίσης ελέγχει τη σωστή ρύθμιση της θέρμανσης και την σωστή χρήση της ενέργειας επομένως. Άρα θα ήταν ενδιαφέρον να δει κανείς το θέμα και από την άποψη αυτή. Εάν δηλαδή τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν πλέον τις ικανότητες και τα προσόντα αυτά. Και εκεί ποιος θα ήταν ο ρόλος τους και ποιες θα είναι οι ελλείψεις που θα προκύψουν εκ των υστέρων εφόσον αντικαταθούν από άλλα πρόσωπα με λιγότερα επαγγελματικά προσόντα. Επίσης η διατάξεις, οι οικοδομικές διατάξεις που και εκεί μάλιστα διαφέρουν από ε, καντόνι σε καντόνι. Και τίθεται και θέματα πώς ε, προστατεύονται τα υπόγεια νερά και πώς προστατεύονται οι γείτονε σε περιπτώσεις ε, οικοδομικών εργασιών. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη και τότε νομίζω ότι αυτές οι ελλείψεις που διαπιστώνεται θα φωτιστούν από τελείως διαφορετικό φως. πολύ ενδιαφέρουσε πληροφορίε. Το ερώτημα είναι εάν υπάρχουν διακρίσεις ε, για λόγους εθνικότητας και όχι εάν είναι τα προσόντα, εφόσον έχουν τα συγκρίσιμα προσόντα βεβαίω, Και Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης για την ενημέρωση, την πολύ χρήσιμη ενημέρωση και χαίρομαι που συνεχίζετε να εργάζεστε για την εφαρμογή της οδηγίας υπηρεσιών, που είναι σημαντικό τμήμα της εργασίας του Ευρωκοινοβουλίου. Και εμείς οι Ευρωβουλευτές βέβαια είχαμε συμβάλει τότε να είναι λογική και η τελική μορφή που δόθηκε, έχοντας αφαιρέσει την αρχή της χώρας προέλευσης και με τον τρόπο αυτό ευνοώντας το άνοιγμα των αγορών ώστε να υπάρχουν κανόνες, αλλά οι κανόνες αυτοί να μην σημαίνουν προσκόμματα. Από τις διάφορες παρεμβάσεις προκύπτει νομίζω ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η ετερογένεια, όπως την είπε ο κ. Πέκμανς, Αυτή η διαφορετικότητα των δικαιικών πλαισίων σε διάφορες χώρες μέλη. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και που θα ήθελα εγώ να αντιμετωπίσω και το ερώτημα που προκύπτει από αυτό είναι τι σημαίνει αυτό για το μέλλον. Επανέρχομαι σε κάτι που είπε και ο Σπέλκμανς. Ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα απορρίθμιση, αλλά μάλλον δημιουργία κοινού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να καταργηθεί αυτή η ετερογένεια. Εκεί θα ήθελα να θέσω μερικά ερωτήματα και προς όλους τους ειδικού. Γιατί αυτό νομίζω ότι είναι το ουσιώδες αυτά που ακούσαμε. Αλλά έχω και μια ειδική ερώτηση για τον κύριο Πέλκμανς. Λέτε στη σελίδα 14 να διακρίνεται η διοικητική ετερογένεια από την πραγματική διαφορετικότητα. μπορείτε να εξηγήσετε τι ακριβώς εννοείτε. Μου φαίνεται σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι ωραία και πομπόδης κάπως η φράση αυτή, αλλά δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη για μένα και γι' αυτό να μου την εξηγήσετε. Και εμείς ζητήσαμε εξ αρχής να μας δώσετε και ωραία σαφή συγκεκριμένα παραδείγματα. Γι' αυτό δεν μου αρέσουν τόσο πολύ αυτές οι ωραίες και μεγαλόσχημες φράσεις. και κάπως ε, με έχει δυσαρέστησε κάτι που είπε η κυρία Κοράτσα Μπίλτ, η οποία αντίπε στην κυρία Νίλσεν που μίλησε για την οδηγία απόσπαση εργαζομένων. Εάν σα ενοχλεί που δεν μιλούμε μονάχα για την οδηγία υπηρεσιών, τότε θα έπρεπε ήδη να παρέμβετε όταν μίλησε ο κύριο Πέλκμανς ή η κυρία Όμεν, που αναφέρθηκαν και σε άλλε οδηγίε, μεταξύ άλλων στην οδηγία για την αναγνώριση των προσόντων. Είτε λοιπόν μπορούν όλοι να αναφέρονται και σε άλλε οδηγίε, είτε κανένα. Αυτό α το πούμε από την αρχή, ώστε να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση των ομιλητών. Ο κύριος Πέρμαν ήταν πολύ σαφής ε, για ολόκληρη αυτή τη δέσμη οδηγιών που αφορούν ε, την οδηγία υπηρεσιών. Και κυρία Ράπτη βεβαίως στη συνέχεια μετά την κυρία Χάνσλικ. Συγγνώμη, ε, κατόπιν ετήματος κυρία Σαράπτη θα ε, λάβω και εγώ το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερως που και πάλι ασχολούμαστε με την ε, οδηγία υπηρεσιών και εγώ ασχολήθηκα με αυτό κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και είχα προσκαλέσει τον Πολωνό υδραυλικό σύμβολο του συμβιβασμού ε, που είχε ολοκληρωθεί με την σύμβαση της οδηγίας περιπηρεσιών και γι' αυτό με τα χαράς ε, και με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να τονίσω ότι ε, δεν είμαι ικανοποιημένη με τη λειτουργία της οδηγίας υπηρεσιών στην ενιαία αγορά. έχει αρχίσει να εφαρμόζεται μόνο τρία χρόνια τώρα. Υπάρχουν κάποια διοικητικά εμπόδια και φραγμοί που αναφέρθηκαν σήμερα και αυτό σημαίνει ότι η παροχή αυτών των υπηρεσιών είναι εξαιρετικά δύσκολη και τα στατικά στοιχεία μας δείχνουν ότι όταν υπάρχει η άρση των φραγμών, αν υπήρχε μάλλον η άρση των φραγμών, η παροχή των υπηρεσιών θα ήταν μακράν καλύτερη. δεν ξέρω αν θυμάστε τότε που μας είχαν δοθεί κάποια στοιχεία το Δανικό Ινστιτούτο, ότι αν εφαρμοζόταν κατάλληλα η οδηγία, τότε 1,5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στην Ευρώπη. Και 1,5 εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας, λοιπόν, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν αν εφαρμόζαμε σωστά την οδηγία και αν ε, μπορούσαμε να οδηγήσουμε στην άρση των φραγμών. Τώρα, να επικεντρωθώ στα όσα είπε η κυρία Νίλσεν. Εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας ε, του ΕΛΚ είμαι και σκιώδης εισηγήτρια και δεν μπορώ να συμφωνήσω με τα όσα είπατε κυρία Νίλσεν. Οι προτάσεις σας, κατά τη γνώμη μου, ουσιαστικά οδηγούν σε περαιτέρω προστατευτισμό για τον εργαζόμενο. Βέβαια, εγώ διαφωνώ με την προστασία του εργαζομένου, αλλά όταν μιλάμε για την απόσπαση εργαζομένων, ε, η επιχείρηση δεν μπορεί κατά την απόσπαση να ε, επιβαρύνεται με υπερβολικό άχθος. Αναφερθήκατε και στην κρίση και στο πώς μπορούμε να ξεφύγουμε. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια ισορροπία εδώ. Να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 4, εκατομμύρια και νέες θέσεις εργασίας. Πρέπει να βρεθούν οι άνθρωποι που θα τις αναλάβουν λοιπόν. Και οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Στα άρθρα 3 και 9 είναι εντελώ διαφορετικό από αυτό που είπε η κυρία Νίλσον. Βεβαίω και, στα, και στο άρθρο 3 θα έχουμε ανοιχτό κατάλογο στο άρθρο 9, κλειστό κατάλογο και στο άρθρο 12. Δεν θέλουμε να έχουμε ε, αυτή την ευθύνη, το liability. Θα δούμε τι θα γίνει με την ε, ψηφοφορία, αλλά ας προσπαθήσουμε να επιτύχουμε την κατάλληλη ισορροπία που θέλουμε να επιτύχουμε για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζομένους. Σίγουρα εκτός ε, πεδίου εφαρμογή και αντικειμένου, αλλά δεν πειράζει και πάλι με ποιικής. Είδα στη συνέχεια ότι η της Λιμπερασιών λέει σήμερα η ε- Ευρώπη μετά ε, τον ε, Πολωνό Ιδραυλικό, ο, Άγγλ, ο Άγγλος εκπαιδευτής σκι. Κυρία Στάιλερ, έχετε το λόγο. Yes, ma. Ευχαριστώ. Και βεβαίως μπορείς να έρθεις στη Σκωτία όποτε θέλεις να κάνεις σκι, Πρόεδρε. Τώρα, λίγο πιο σοβαρά για την υλοποίηση και την ισορροπία. Σίγουρα είναι εύλογα αυτά τα στοιχεία, όμως πρέπει να εξετάσουμε στοιχεία από τις δικής μου τουλάχιστον πολιτικής ομάδας αφορούν ε, τις ε, απόσπες εργαζομένων έχουμε 24 εκατομμύρια ανέργους αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί από αυτούς είναι νέοι άνθρωποι. Μιλάμε για ανάπτυξη, θέσεις εργασίας. Βεβαίως και οι υπηρεσίες είναι πολύ σημαντικές σε αυτό το τομέα. Πρέπει να δούμε πώς βρίσκουμε λοιπόν αυτή την ισορροπία και στην ανάπτυξη και στην κοινωνική προστασία. Και είδα κάτι πριν στο Business Europe νομίζω, κάτι που με απασχόλησε λίγο για αυτή την μηδενική ασφάλιση. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες διευκρινήσεις πού ακριβώς αναφερόσασταν. Γιατί τελικά όλοι έχουμε τους ίδιους ε, στόχους. Έχουμε αυτό το πολύ, την πολύ ωραία φύσα, το lift off, δηλαδή την ε, απογείωση για τις θέσεις εργασίας, την απασχόληση. Σίγουρα το θέλουμε όλοι αυτό, αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν και τα κατάλληλα επίπεδα προστασίας. Να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα στη δική μου εκλογική περιφέρεια. Είχαμε μια πολύ επιτυχή επιχείρηση υπηρεσιών που μέσα στα Χριστούγεννα ε, πήγαν κάτω στο κατάλογο, έδωσαν έναν ε, κατάλογο εργαζομένων και αυτοί οι άνθρωποι κατευθείαν απολύθηκαν, τους έδιωξαν από τις εγκαταστάσεις και δεν μπορούσαν καν να μπουν μέσα στο, ε, στο πάρκινγκ του καταστήματος και έπρεπε να περιμένουν κάποιον εκεί έξω να έρθει να τους πάρει. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα κακομεταχείριση εργαζομένων και μάλιστα ε, πολλές φορές ε, υπάρχουν και πολλές κακές ε, απολαβές. Στον Ηνωμένο Βασίλειο, στην πλειοψηφία των φτωχών οικογενειών, ένα μέλος οικογένειας απασχολείται. Έτσι έχουμε πολλαπλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε και είναι σημαντικό να θίξουμε και αυτά τα κοινωνικά ζητήματα. Όμως θεωρώ ότι οι υπηρεσίε είναι σημαντικές, είναι ο παράγοντας ανάπτυξης της ε, οικονομίας μας. Έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε σωστά και ε, ευχαριστώ τους ομιλητές που ήρθαν εδώ. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους των συναδέλφων που είμαστε τόσο λίγοι εδώ σήμερα. Θα πρέπει να ε, καλούμε και τους ε, συναδέλφους μας, υπόλοιπους ευρωβουλευτές, να παρευρίσκονται πιο συχνά σε τέτοιου είδους συνεδριάσεις, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικές. Ευχαριστώ όλους τους μιλητές για τις προσπαθίες τους. Thank you very much. Well, Ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο σύντομα ερωτήματα και μετά θα δώσω το λόγο ε, στο πάνελ. Αλλά ας το αντιστρέψω τη σειρά, μετά θα ξεκινήσω πρώτα από την κυρία Νίλσεν. Ελπίζω να τα καλύψετε όλα τα σημεία, αλλιώ εγώ θα σα τα επενθυμίσω. Να επιστρέψουμε σε αυτό που μα απασχολεί σήμερα. Η δημιουργία ευκαιριών και θέσεων εργασία. Κατανοώ ότι όλα τα ζητήματα ε, αυτά στην οδηγία υπηρεσιών σίγουρα μας απασχολούν σε ό,τι αφορά την απόσπαση εργαζομένων και πώς θα επιλύσουμε τέτοια ζητήματα. Η Επιτροπή ε, έκανε μια άμεση παρέμβαση για τη διευκρίνηση των διατάξεων αυτής της οδηγίας. Υπήρχαν πολλά ζητήματα λοιπόν εκεί, όμως ε, πράγματι η επιβολή ε, των, ε, της νομοθεσίας δεν έχει σχέση με αυτή την ε, οδηγία. Και η κυρία Νίλσον έχει δίκιο ότι μιλάμε για την επιβολή των ε, κανόνων της ενιαίας αγοράς, αλλά προφανώς υπάρχει τεράστια διαφορά και πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες οδηγίες ε, του δικαίου απασχόλησης της εργατικής νομοθεσίας. Αλλά δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε αυτά τα δύο εδώ, τις δύο οδηγίες. Για τα όσα ε, είπαν οι συνάδελφοι, για αυτή την έλλειψη ομοιομορφίας, αυτή την ετερογένεια, ιδιαίτερα ακαδημαϊκός όρος, εγώ προσπαθώ να βρω έναν πιο απλό. Εγώ διερωτώ με μήπως θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στην επιβολή αντί για τις ε, δυνατότητες. Πρέπει να δούμε στο βαθμό, το βαθμό στον οποίο έχουν αρθεί κάποιοι φραγμοί σε ορισμένες οικονομίες. Αυτό προκαλεί εντύπωση, για παράδειγμα, είναι ότι η Ισπανία έχει επιτύχει υψηλά επίπεδα άρσης ή μείωσης τέτοιων φραγμών. Και βεβαίως ποια οικονομία αυτή τη στιγμή χρειάζεται περισσότερες θέσεις εργασίας. Σίγουρα η μείωση τετοιων φραγμων και βεβαιως ποια οικονομια αυτη τη στιγμη χρειαζεται περισσοτερες θεσεις εργασιας σιγουρα η ισπανια αν λάβουμε υπόψη και το μέγεθος της οικονομίας. Πρέπει λοιπόν να δούμε ε, αυτά τα στοιχεία, ε, το μέγεθος και τις οικονομικές δυνατότητες. Και τότε ούτε η Γερμανία τα πάει πολύ καλά, γιατί είχε μικρότερη μείωση φραγμών. Ξέρουμε βέβαια ότι είναι μια εξαιρετικά ισχυρή οικονομία. Ίσως πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτές, αυτούς τους δείκτες και να δούμε πού ακριβώς υπάρχει το αναξιοποίητο δυναμικό. Εκεί ίσως θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερες θέσεις εργασίας. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το, την ε, σημασία του επαγγέλματο του καπνοκαθαριστή που ανέφερε ο Αυστριακό συνάδελφο και πώ πρέπει να ενθαρρύνουμε τον κόσμο, κατά πόσο πρέπει να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να έχει ε, άλλου είδου θέρμανση και το καθεξή στο σπίτι του. Ε, σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα όμω, ε, η Αυστρία είναι πολύ χαμηλά στον κατάλογο θα μπορούσε να τα πάει πολύ καλύτερα αν είχε αυξήσει την παραγωγικότητά της με την εφαρμογή της ε, οδηγίας περιπηρεσιών. Αυτά ήθελα να πω. Ξαλάφρωσα τώρα η κυρία Νίλσον. Έχετε ένα-δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω από το πρώτο ερώτημα τι περιμένουμε ως αποτέλεσμα της πρότασης για περαιτέρω απελευθέρωση. Όταν πρωτοσυντούσαμε αυτή την οδηγία πριν από χρόνια, η θέση μας ήταν ότι θα πρέπει πόσε υπηρεσίες να είναι εκτός. Όχι, με συγχωρείτε, ο πρόεδρος, να είστε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Κοιτάξτε μένα, άμα σας δυσκολεύει, για να βλέπετε και το μικρόφωνο. Λοιπόν, η θέση μας αυτής εξ αρχής ήταν ότι δεν θέλουμε να συμπεριληφθούν και οι δημόσιες υπηρεσίες στην οδηγία. Γιατί η απελευθέρωση θα οδηγήσει σε κακές υπηρεσίες και κακές συνθήκες εργασίας, κακούς μισθούς. Ήδη έχουν γίνει μελέτες που στο Ηνωμένο Βασίλειο είδαμε τα αποτελέσματα ιδιωτικοποίησης δημόσιων υπηρεσιών και για τις υπηρεσίες αλλά και για τους εργαζομένους που δουλεύουν σε ε, ιδιωτικές εταιρείε πλέον. Βεβαίω η μελέτη αφορούσε του χαμηλότερου μισθού, αλλά ήταν σαφέ ότι ήταν και χειρότερε υπηρεσίε που παρήχαν πλέον. Για το ερώτημα τη κυρία Κεπάρτ. Για μα. το μείζον είναι η οδηγία για τι υπηρεσίε και το δικαίωμα ελευθερία εγκατάσταση θα μην είναι αντικείμενο κατάχρηση και παραβίαση τη εθνική νομοθεσία για τα εργασιακά. Για μένα η σύνδεση είναι προφανής. Μιλάμε για τι ασυνοριακέ υπηρεσίες. Αποσπώνται εργαζομένοι για να κάνουν διασυνοριακά μια εργασία. Ε, δεν είναι κάτι διαφορετικό, αλλά δεν μπορούμε να, να, μιλάμε χωριστά για τα θέματα ε, τα εργασιακά, παρά μόνο και μέσα σε αυτό το ζήτημα. Δεν απαντήσατε όμως το ερώτημά μου για την εφαρμογή. Θα μου απαντήσετε αργότερα. Ποιες χώρες πρέπει να τα πάνε καλύτερα. Ναι, ναι να απαντήσω. το συγγνώμη, το ξέχασα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο κύριος Μάρι. Εγώ εδώ δεν μιλώ εξ ονοματός μου, ούτε καν εξ ονόματος της Ιρλανδικής Αντιπροσωπείας. Προσπαθώ να σας παρουσιάσω α, κάποια αποτελέσματα από τη συζητήσεις στο Συμβούλιο και τις θέσεις των Υπουργών και των κρατών μελών. Να το διευκρινίσω αυτό πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, να μιλήσαμε και για άλλες οδηγίες που συνδέονται με τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία, συνθήκες εργασίας κτλ. Όλα αυτά συνδέονται με την οδηγία της υπηρεσίας. Οι συνάδελφοι στην Προεδρία που προείσταται αυτών των εξειδικευμένων ομάδων εργασία συμμετέχουν στους τριμερείς διαλόγους με το Κοινοβούλιο. Οπότε φαντάζομαι ότι θα γίνει κάθε προσπάθεια για ισορροπημένες λύσεις που να ικανοποιούν όλους. Ελπίζω αυτά να γίνουν κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας. Όλες οι αναφορές ε, για τα παραδείγματα του Πολωνού Ιδραλικού Τυπέρναν και αναλογίες ακούστηκαν, αλλά το, η όλη συζήτηση για τα κατοχυρωμένα ε, επαγγέλματα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι ε, έχει γίνει, αλλά θα πρέπει να γίνει και μια ουσιαστική συζήτηση για όλα τα επαγγέλματα και να συνεχίσει η συζήτηση στο Συμβούλιο, ειδικά γι' αυτό. Η εφαρμογή της οδηγίας της είναι κάτι που γίνεται βαθμία, που μπορεί να γίνει βαθμία. Είναι μια διαδικασία Άρα σε νομικό επίπεδο είναι μια διαδικασία και υποστηρίζουμε ως Προεδρία τη διαδικασία screening που γίνεται το διάλογο μεταξύ ομοντήμων, το peer review δηλαδή. Όλα αυτά τα στηρίζουμε. Ε, η σύσταση μια άλλη ομάδα υψηλού επίπεδου είναι καλό να γίνει το στομότερο δυνατόν. Οι οδηγίε τη υπηρεσία θα ενταχθεί στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Και άρα στο μέλλον θα υπάρχουν και συστάσεις που θα απευθύνονται σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη, με συγκεκριμένους στόχους εφαρμογής και θα υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις που θα πρέπει να φέρουν εις πέρας ε, τα κράτη-μέλη. Ας περιμένουμε λοιπόν λιγάκι με τις καλοκαιρινές διακοπές, το φθινόπωρο, να δούμε τις συστάσεις της Κομισιόν και πού θα καταλήξει το Συμβούλιο μάλλον ε, πιο σκληρά θα είναι τα πράγματα, πιο πολύ μαστί και το θα ε, βλέπουμε στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα, τι είναι το μείζον, ποιο είναι το, το σημαντικότερο. Αυτό που προσυπογράψαμε είναι να εφαρμόσουμε και να επιτύχουμε τους ε, απότερους σκοπούς αυτής της οδηγίας. Από ό,τι γνωρίζω, δεν υπάρχει κάποια πρόταση στο τραπέζι για περαιτέρω απελευθέρωση των υπηρεσιών. Τουλάχιστον δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα της Προεδρίας. Αν απαιτείται περισσότερη νομοθεσία για την καλύτερη εφαρμογή της κείμενης οδηγίας, εντάξει. Και αν απαιτηθούν διαδικασίες παράβασης, ας υπάρξουν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρία Σούμερ. Όμερ, συγγνώμη. Ναι, να απαντήσω πρώτα απ' όλα στο ερώτημα της κυρίας Ράπτη για το άρθρο 20 και την α, υπηρεσίες, την πρόσβαση υπηρεσίες. Πρώτα απ' όλα, οι της επιχειρήσεις υπηρεσιών είναι προς συμφέρον τους να μην έχουν διαφορετική αντιμετώπιση, γιατί και οι ίδιες επιχειρήσεις είναι πελάτες άλλων επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες. Υπάρχουν βεβαίως κάποια αντικειμενικοί λόγοι για κάποια διαφοροποίηση στη μεταχείριση. Να είμαστε προσεκτικοί. Να μην δίνουμε υπερβολικό βάρος στις επιχειρήσεις. Ένα σύντομο παράδειγμα. Μια μικρομεσαία επιχείρηση στις νότιες κάτω χώρας, που πρέπει να κατασκευάσει ένα ποδήλατο για μια μακρινή χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αναλογικό να ζητήσει από αυτή την εταιρεία να κάνει μια έρευνα για το πώς θα πρέπει αυτό το ποδήλατο να κατασκευαστεί καλύτερα, 500 χιλιόμετρα μακρύτερα, γιατί θα είναι προς όφελος του καταναλωτή. Δηλαδή αυτό μπορεί να το κάνει συμφέρει μια μικρομεσαία επιχείρηση. Πρέπει να ε, πούμε μεν ότι κατά λοιπά δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση ούτε στις τιμές, εκτός από κάποιους αντικειμενικούς λόγους. Αυτό θα απαντούσα στο ερώτημά σας. να απαντήσω στον κύριο Λόκαρτ. Γιατί πρόοδο έχουμε κάνει ως τώρα. Μα φυσικά έχει γίνει πρόοδος και φυσικά συγχαίρουμε τα κρατημέλη για την πρόοδο που έχουν επιτύχει. Αλλά λείπουν και άλλα πράγματα που δεν έχουν γίνει. Μου ζήτησε τα παραδείγματα. Ήδη ανέφερα κάποια αλλά παρατηρούμε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που χρειάζονται διπλές άδειες με το που αλλάζουν χώρα δραστηριότητας. Υπάρχουν ε, λοιπόν υπερβολικές απαιτήσει για τις άδειες, για τις μεταφράσεις, ε, πολλά τέτοια παραδείγματα. Και σίγουρα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτές οι επιχειρήσεις είναι τι περιθώριο λιγμού έχουν σε ό,τι αφορά την αρχή της αναλογικότητας. Ελπίζω να σας απαντώ. Και ο κύριος Πέλμαν τέλος. Ευχαριστώ. Τέσσερα θέματα θέσατε σε μένα, αν κατάλαβα καλά. Ιδίω για του αποσπασμένους. Ξέρετε, ε, εγώ είμαι αναφανών υπέρ των αποσπασμένων, αλλά όχι, δεν είμαι υπέρ τη οδηγίας. Γιατί η οδηγία επιτρέπει την κατάχρηση και πολύ κακές καταστάσεις. Για πολλούς λόγους, λοιπόν, θα πρέπει να εξαφανιστεί αυτή η οδηγία. Οπότε να έχουμε προσωρινές, βραχίδιες, διασυνοριακές υπηρεσίες, τις οποίες να σεβόμαστε, να σεβόμαστε τους κανόνες. Γιατί? Ένας λόγος για τους οποίους εγώ θέλω να επισημάνω, για τους τηρώνται λιγότερο η όροι, είναι ότι υπάρχουν τρεις χώρες στην Ένωση που δεν έχουν νομοθεσία περί κατώτατου μισθού. Εκπληκτικό αυτό προσπάθησα με κάθε γενναιότητα ως οικονομολόγος να διτείνω στους Γερμανούς οικονομολόγους που είναι κατά να, να με εξηγήσουν γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα. Το ίδιο στη Σουηδία και τη Δανία. Η Σουηδία όχι ακόμα, αλλά στη Δανία σε μια μεγάλη διάσκεψη του έλεγα «Μα πώς είναι δυνατό να μην έχετε νομοθεσία περί κατώτε του μισθού». Μια σελίδα να είναι αυτός ο νόμος. Και δεν λέω ότι μετά με τι τη υπηρεσίε και για του αποσπασμένου εργαζόμενου θα έχουμε λύσει όλα, τουλάχιστον θα έχουμε πολύ λιγότερα προβλήματα. Δεν μπορούμε δίπλα στη Γερμανία να έχουμε την Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία που δεν έχουν κανένα τέτοιο πρόβλημα γιατί υπάρχει η νομοθεσία κατά το κατώτατο μισθό. Δεύτερο σχόλιο για την Αυστρία. Μπορεί να μην με πιστεύετε, αλλά ξέρετε τι συνέβη. Χθε εμά μα καθαρίσανε την καμινάδα. Δεν ήταν αυστριακό όμω ο λειτουργό. Εντάξει, μη συγγνώμη. Εγώ τον πλήρωσα προσωπικά. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό με τις καμιναδές στην Αυστρία. Λόγω της ασφάλειας. Χρειάζεται επαγγελματικό καθαρισμό για να μπορεί να υπάρχει ασφάλεια στι κατοικίε. Υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμό και είναι καλό αυτό. Αλλά δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν για δεκάρες, για πενταροδεκάρες. Νομίζω ότι αν τα δούμε τα πράγματα σωστά, αυτό είναι υπέρ του ανταγωνισμού. Άρα λοιπόν όλα δείχνουν στο, υπό το πρίσμα της αναλογικότητας. Και για τους καθαριστές καμινάδες και Βλέπω σε πολλές περιπτώσεις το θέμα της αναλογικότητας, τουλάχιστον εγώ. Πρώτα απ' όλα, το απόλυτο είναι αυτό αναγκαίο. Το δικαστήριο αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα με αυτό το θέμα. Το άλλο όμως ζητήμα είναι το πλέον προφανές. Ο Επιτροπός Μπαρνέ πολύ συχνά τι άκουγε, ξέρω να πας στη Γερμανία να πας να τους πεις ότι δεν πρέπει να τύχαν προστασία σε όλα, αυτά τα τόσο σημαντικά α, επαγγέλματα. ας αφήσουν να το λύσουν αυτά τα κράτη-μέλη. Ξέρετε, μεταξύ των κράτη-μέλη μπορούν να τα λύσουν μεταξύ τους πολύ εύκολα. Δηλαδή δεν μπορεί 24 να το κάνουν με έναν τρόπο και άλλοι τρει διαφορετικά. Εξηγήστε μας εσείς οι τρεις πώς βλέπετε το σωστό και εμείς δεν το βλέπουμε. ελπίζω, ελπίζω να μπορέσουμε να άρουμε σε μεγάλο βαθμό όλου του περιορισμού, αν τα δούμε τα πράγματα από την σωστή οπτική γωνία. Κυρία Κεφχάρτ, τη σέβομαι ιδιαίτερα. Ήταν συγγήτρια ε, πριν από τρία χρόνια για ένα θέμα από το που είχε γύρει πάρα πολύ την συζητήσει, ίσω πιο έντονο εκτό από το θέμα του Ρίτ. Σε εγώ δεν υπονόησα πουθενά την απορρίθμιση, την απελευθέρωση. Τίποτα ε, τέτοιο δεν διαφάνισε σε διαφάνειές μου. Εκτός ε, αν κάπου είναι απαραίτητο. Ούτε αυτό εννοούσαμε την ετερογένεια. Ούτε μιλάμε για απόλυτη διαφορετικότητα. Αν ένα κράτος μέλος έχει μια συγκεκριμένη προτίμηση, θα πρέπει να υπάρχουν και σαφή επιχειρήματα υπέρ αυτή. Αλλά η ετερογένεια τι είναι. Πού οφείλεται μάλλον. Στη γραφειοκρατία, στους εφαρμοστικούς νόμους, στο ότι Απλό καθένας καθένα έχει επιλέξει να το κάνει με διαφορετικό τρόπο. Τεχνικοί ε, μηχανισμοί και όλα αυτά οδηγούν στην ετερογένεια. Άρα θα πρέπει να ερευνήσει πώ. Πα στη βάση δεδομένων του ΩΣΑ. Δεν πρέπει να το κάνετε τώρα, γιατί είναι φρικτή δουλειά. Αλλά αν το κάνετε θα δείτε με τα μάτια σας τα 30 μέλη του ΩΣΑ, που είναι και τα πιο πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης, 23 κράτη-μέλη ε, της Ένωσης είναι στον ΩΣΑ, σε πολλά στοιχεία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν διαφορές. Και εκεί είναι που πάσχουμε. Εγώ δεν είπα ότι θα πρέπει αυτά να τα <laughs> διαγράψουμε όλα και να επιβάλλουμε κάτι ενιαίο από πάνω. Απλά λέμε ότι η εναρμόνιση δεν είναι αναγκαστικά κάτι κακό, κάτι που επιβάλλεται. Μπορεί η εναρμόνιση να γίνει και θελοντικά. Να δώσω ένα παράδειγμα του τι κάνουν στις ΗΠΑ. Στις ε, ΗΠΑ, οι Αμερικανικές πολιτείες έχουν πάνω από ε, έχουν πολλές εθελοντικές ενώσεις, combats, όπου συζητούν θέματα εναρμόνισης. Πράγματα τα οποία δεν απαραίτητο να ρυθμιστούν μέσω της νομοθεσίας, αλλά ε, δημιουργούν αγκάθια ε, στο εμπόριο. Δεν υπάρχει όμως ποντιακή νομοθεσία για αυτά τα ζητήματα. Αυτού του είδου λοιπόν οι ενώσει, αυτά τα κόμματα έχουν στι ΗΠΑ, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ είναι ομάδε που ε, συζητούν αυτά τα θέματα που μπορούν να ε, ευθυγραμμιστούν. Τέλος πρόεδρε, η Ισπανία είναι μία από τι χώρε εκείνες που προέβησαν σε δραστική απελευθέρωση και δεν χρειάζονταν κανένα μόντι. Στην Ιταλία εν μέρει έγινε μέσω του κυρίου Μόντι τα θέματα απελευθέρωση πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα. Ξέρετε, η οδηγία έχει πολύ λίγα χρόνια ζωή. Μιλάμε για αποτελέσματα από το 2009-2010. Σήμερα η Ισπανία σε τέτοια βαθιά κρίση που δεν μπορεί να δει άμεσα θετικά αποτελέσματα. Είναι αδύνατο στη σημερινή κατάσταση και ακόμα και αν υπάρχουν δεν είναι μετρήσιμα στοιχεία. Μακροπρόθεσμα όμως αυτή η απελευθέρωση θα βοηθήσει την Ισπανία. Όταν θα ε, επανέλθει, θα έχουμε την ανάκαμψη, θα δείτε αποτελέσματα. Είναι καλά λοιπόν τα νέα. Και γενικότερα, Πρόεδρε, και κλείνω, στην ε, Μπρίζ προσπαθήσαμε να δούμε με τις σπουδαστέ μας τέσσερις χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιρλανδία και Ελλάδα, η Ιρλανδία δεν είναι τόσο πρόβλημα, πώς αυτά τα προγράμματα που τους έχουν επιβληθεί σε αυτές τις χώρες, έτσι από ότι είναι πιο σκληρά τα πράγματα, κατά πόσον τελικά θα οδηγήσουν σε βαθιές μεταρρυθμίσεις. Απάντηση αν πιστέψετε αυτά που λένε οι εκθέσει, τριμηνέ εκθέσει τη Τρόικα, γιατί δεν σημαίνει ότι αυτά που λένε σε εκθέσει συμβαίνουν κιόλα. Αλλά αν ήταν όλα αυτά αλήθεια, τότε η Ελλάδα θα ήταν σούπερ ανταγωνιστική χώρα σε τρία χρόνια από σήμερα. Ωραία, λέει ο Πρόεδρο. Δεν θέλω να ξεκινήσω τώρα συζήτηση για τον κατώτατο μισθό, αλλά και θα καλέσω του συναδέλφου να τοποθετηθούν αργότερα γι' αυτό. Πρέπει να προχωρήσουμε. Αλλιώς θα έχουμε τελείως εκτός χρόνου. Και αν θέλετε, μπορείτε να τους περιλάβετε και στην απάντησή σας αργότερα. Λοιπόν, πάω στους τρεις επόμενους ομιλητές, γιατί πρέπει να δούμε το θέμα της ε, καινοτομία και τη μεγιστοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων τι επιχειρήσει και του καταναλωτέ. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ράινχολτ Σράτς, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή στην Αυστρία που θα μας μιλήσει για την οπτική γωνία του καταναλωτή. Θα μας μιλήσει ο Φρόνσο Μομπουάς, πρόεδρο της e-commerce Europe για τις προκλήσεις για τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Και τέλος, η κυρία Λένα Γιώχανσον, Γενική Διευθύντρια του σουηδικού PSC που επισκεφτήκαμε πριν κάποια χρόνια και είχαμε εκπλαγεί ιδιαίτερα από την όλη δουλειά που κάνουν οι αρμόδιες σουηδικές αρχές ε, για την αδειοδότηση των παρόχων υπηρεσιών. Θα είμαι πιο αυστηρό με το χρόνο αυτή τη φορά. Δεν ήμουν πολύ βεβαίω και πριν. Τέλο πάντων, έχετε το λόγο κύριε Σράντ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, Κυρία Συγήτρια και αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να σας μιλήσω για την οδηγία υπηρεσιών και την σχέση που έχει με τους καταναλωτές. Με απασχολεί κυρίως το άρθρο 20 παράγραφος 2, γιατί λάβαμε πολλές καταγγελίες από καταναλωτές σχετικά με αυτό. Για όσους εξημών, παρακαλώ τη διαφάνεια. Να συνεχίσω να μιλώ ή να περιμένω. Καλά, συνεχίζω τότε. Για όσους εξημών δεν γνωρίζετε το άρθρο 20 παράγραφος 2, αυτό απαγορεύει τη διακριτική μεταχείριση στην βάση εθνικότητας ή τόπου κατοικίας από πλευράς παρόχων υπηρεσιών. Διαφορετική μεταχείριση επιτρέπεται μόνο εφόσον αιτιολογείται από αντικειμενικά κριτήρια. Όταν κανείς αναφέρεται στο 20 παράγραφος 2, εννοεί επίσης και τους σχετικούς εθνικούς εφαρμοστικούς νόμους. Πώς λοιπόν τη το ερώτημα μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές δεν θα γίνουν θύματα διακρίσεων βάσει του τόπου ε, ε, κατοικίας τους ή της εθνικότητάς τους. Πρέπει πρώτα να ευαισθητοποιηθούν οι καταναλωτές. Επίσης να υπάρχει βοήθεια από τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών. Επιβολή του νόμου και ενίσχυση της συνεργασίας με τις αρχές ανταγωνισμού. Αν ίσως μπορείτε να προχωρήσετε τις διαφάνειες. Πολύ ωραία το επόμενο τότε, η επόμενη διαφάνεια, πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα να αυξηθεί η ευαισθησία, να ευαισθητοποιηθούν δηλαδή οι καταναλωτές. Εμείς το βλέπουμε καθημερινά αυτό. Δεν γνωρίζουν οι καταναλωτές περί της οδηγίας. Ή δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή απαγόρευση. Συχνά αποδέχονται τις διακρίσεις λόγω του ότι δεν γνωρίζουν ότι απαγορεύονται. Εκεί πρέπει να παρέμβουν τα κέντρα καταναλωτών. Και εμείς τώρα επεξεργαζόμαστε μια κοινή θέση για να ενημερώνουμε τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους και ιδίως αυτά που απορρέουν από το άθρο, 2, από το, ε, 20 παράγραφος 2. Έχω και παρόντα συναδελφό μου από το ICCL, από άλλο ε, το όργανό μας δηλαδή. Γιατί όμως αυτή η ευαισθητοποίηση είναι τόσο σημαντική. Εφόσον γνωρίζουν τα δικαιώματά του οι καταναλωτέ, μπορούν να επιμείνουν στην παροχή τη υπηρεσία εφόσον αντιμετωπίσουν αδικαιολόγητη άρνηση. Επόμενη διαφάνεια σα παρακαλώ. Η βοήθεια, η υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών. Υπάρχουν περιπτώσει που δεν μπορούν να επιλύσουν οι καταναλωτέ μόνοι του εκεί μπορούν να βοηθήσουν τα κέντρα καταναλωτών. Γράφουμε στους ε, παρόχους υπηρεσιών και συχνά ε, πετυχαίνουμε λύσεις. Γιατί η κοπελίτσα από την Χαβάη θα με ρωτήσετε το, το σχεδιάκι αυτό. Ένας αυστριακός καταναλωτής ήθελε να νοικιάσει, να ε, κλείσει ένα αυτοκίνητο ενοικιαζόμενο δηλαδή στη Χαβάη για τις διακοπές του γιατί ήταν πολύ φθηνότερο εκεί από ότι στο αυστριακό site. Και την εξοικονόμηση αυτή ήθελε να τη χρησιμοποιήσει η ε, τουρίστη αυτή δηλαδή για να κάνει ένα φούλα φούλα στην ε, ίδια τη Χαβάη. Όμως ο πάροχος υπηρεσιών αρνήθηκε και είπε ότι η προσφορά που είχε στην ιστοσελίδα του ήταν μοναχά για κάτοικους Γερμανίας. Εμείς του γράψαμε, τελικώς το δέχτηκε, αλλά δεν άλλαξε την επιχειρηματική πρακτική του. Πάντως, η τουρίστρια μπόρεσε για κάνει το μάθημα χούλα-χούλα στην Χαβάη. Μου φάνηκε αστείο το περιστατικό και επειδή μου το διήθηκε η ίδια η καταναλώτρια αυτή και γι' αυτό σα το αναφέρω. Να λοιπόν ένα παράδειγμα που μπορέσαμε να επιτύχουμε λύση υπέρ μια συγκεκριμένη καταναλώτρια, όμω ο ε, έμπορο, ο ο πάροχος υπηρεσιών δεν άλλαξε επιχειρηματική πρακτική. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις όπου οι επιχειρηματίες αλλάζουν την, τις πρακτικές τους μετά από τις παρεμβάσεις των κέντρων καταναλωτών και θα σας δώσω ένα παράδειγμα στο επόμενο ε, slide. Οι κουραζιέρες. Μια αυθιακή οικογένεια ήθελε να κρίσει μια κουραζιέρα σε γερμανική ιστοσελίδα για, ε, μιας εταιρείας εγκατεστημένη στην Ιταλία για ένα ποσό 849 ευρώ. ευρώ. Ωστόσο, η εταιρεία απέρριψε την κράτηση αυτή γιατί δεν είχε η οικογένεια ε, τόπο κατοικία στη Γερμανία και τους έστειλε στο αυστριακό, στην αυστριακή ιστοσελίδα. Για την ίδια κράτηση ήταν 2.400 ευρώ. Δηλαδή 1.600 ευρώ και παραπάνω διαφορά η αυστριακή οικογένεια δεν πίστευε στα μάτια της. Δεν πίστευε τόσο μεγάλη διαφορά τιμή, Γιατί άραγε. Και ρώτησε την εταιρεία. Η εταιρεία Κρουαζιέρας τους απίτησε ότι είναι διαφορετική η οικονομική και η κοινωνική κατάσταση στη Γερμανία και στην Αυστρία. Εμείς δεν το πιστέψαμε αυτό, διότι η κοινωνική και η οικονομική κατάσταση στις δύο χώρες για μας είναι πολύ παρόμοια. Ωστόσο η οικογένεια εξακολουθούσε να μην μπορεί να πιστέψει τα πράγματα αυτά και έκανε μια δεύτερη προσπάθεια. Έγραψαν λοιπόν στους travel agents στη Γερμανία, οι οποίοι επίσης απέρριψαν την κράτηση αυτή, διότι τους είπαν ότι το απαγορεύει η εταιρεία της κρουαζιέρας. Απογοητευμένοι λοιπόν οι άνθρωποι ήρθαν σε εμά στο ICC Austria για να τους βοηθήσουμε. Το συζητήσαμε με τους Ιταλούς και γράψαμε τελικά, με το κέντρο καταναλωτών δηλαδή της Ιταλίας, Βλέπετε εδώ τους καινούς καταναλωτές πόσο απογοητευμένοι είναι. Οι Γερμανοί είναι πάνω στο καράβι, ενώ οι Αυστριακοί ε, έχουν μείνει στην αποβάθρα. Μεγάλη απογοήτευση λοιπόν για τα πρόσωπα αυτά. Γράψαμε στην επιχείρηση και η επιχείρηση απάντησε ότι ποτέ δεν θέλησαν να κάνουν διακρίσεις σε βάρος καταναλωτών και ότι από τον Νοέμβριο 2012 και μετά Αυστριακοί αλλά και Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να κλείνουν τις κουραζιέρες τους και στη γερμανική αγορά με τις χαμηλότερες τιμές. Να λοιπόν ένα καλό παράδειγμα που μια μεγάλη επιχείρηση άλλαξε την πρακτική της ώστε να προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά νομοθετήματα και ελπίζω να δούμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, επιβολή. Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις οι οποίες παραμένουν ανεπίδητες. Περιπτώσεις όπου οι έμποροι, οι πάροχοι υπηρεσιών δεν προσαρνούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες και δεν τους αιτιολογούν. Τότε εμείς μεταφέρουμε, τις, ε, διαβάζουμε τις περιπτώσεις αυτές στις αρμόδιες αρχές επιβολής. Μέχρι τώρα όμως το επίπεδο επιβολής είναι πάρα πολύ χαμηλό. Μέχρι τώρα στην Αυστρία δεν γνωρίζω καμιά απόφαση της αρχής επιβολής, αλλά χρειαζόμαστε νομολογία, χρειαζόμαστε αποφάσεις για να ξεκαθαριστούν τα θέματα επιβολής. Ε, οι διάφορες ε, ρήτρε, όροι και συνθήκες της αγοράς. Αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν από τα δικαστήρια. Το Κέντρο Καταναλωτών Αυστρίας απέστειλε ορισμένες από τις υποθέσεις αυτές στις αρμόδιες αρχές, για παράδειγμα με προπληρωμένα τηλέφωνα ή οι ε, ε, κάρτες διαδικτύου στη Γερμανία. Μια γερμανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών αιτιολόγησε την άρνησή της αυτή δεν κάνουν λέει διάκριση διότι ζήτησαν ταχυδρομική διεύθυνση στη Γερμανία και όχι τόπο κατοικίας. Αλλά για μας είναι αυτό το ίδιο. Και η άλλη αιτιολόγηση που πρόβαλε η επιχείρηση είναι το μέγα δίθεν κόστος για να στείλουν τα συμβόλαια στην Αυστρία. Ούτε αυτό το πιστέψαμε, γιατί ζούμε στην ψηφιακή εποχή, ας με το διαδίκτυο. Γι' αυτό το λόγο παραπέμψαμε την υπόθεση αυτή στην αρμόδια αρχή επιβολή στη Γερμανία και αναμένουμε την απόφασή τους. Επίσης τώρα άλλε επιχειρήσεις αυστριακές για αναβατήρες σκι όπου παραπονούνται ορισμένοι ότι πληρώνουν περισσότερα ορισμένοι Ευρωπαίοι από τους ίδιους τους Αυστριακούς. Παραπέμψαμε την υπόθεση στην αρμόδια αρχή στην Αυστρία για να εξεταστεί αυτή η διαφορά τιμών για μας είναι σημαντικό καταναλωτές και από άλλες χώρες μέλη να προσέρχονται στην Αυστρία γιατί έχουμε όμορφα τοπία και ωραίες χιονοδρομικές πίστες και ας έρχονται οι άνθρωποι να τα απολαμβάνουν όχι με υψηλότερες τιμές. Το στείλαμε λοιπόν και αυτό και την υπόθεση αυτή στην αρμόδια αρχή και αναμένουμε την απόφασή της. Επίσης τώρα το δίκαιο ανταγωνισμού. Πολλές από τις υποθέσεις διακρίσεων αποτελούν και παραβιάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού με επιβολή περιορισμών στις πωλήσει στην επικράτεια άλλων χωρών. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να αυξηθεί η συνεργασία με τις αρχές ανταγωνισμού. Παράδειγμα, έλαβα μόλις χθε ένα γνώση να παραδείγματος. Ένας αυστιακός καταναλωτής θέλησε να αγοράσει ένα προκατασκευασμένο σπίτι από μια εταιρεία στην Σλοβενία. Η εταιρεία απέριψε την αγορά αυτή και τον παρέπεμψε στον αυστριακό πολιτή των προκατασκευασμένων σπιτιών λέγοντας ότι έχουν ιδιαίτερη συμφωνία μαζί του και δεν μπορούν να του πουλήσουν απευθεία στο σπίτι. Ο καταναλωτής ήταν πολύ απογοητευμένος διότι η τιμή για ακριβώς το ίδιο προκατασκευασμένο σπίτι ήταν 40.000 ευρώ περισσότερα στην Αυστρία από ό,τι στη Σλοβενία και γι' αυτό ήταν προφανές γιατί ήθελε να το αγοράσει στη Σλοβενία. Η περίπτωση αυτή μας δείχνει ότι πρέπει να συνεργαστούμε με τι αρχέ ανταγωνισμού για να επαληθεύουμε εάν αυτές οι περιπτώσεις ενδεχομένως παραβιάζουν το δίκαιο ανταγωνισμού και ενδεχομένω και το άρθρο 20 παράγραφος 2 της ε, ε, οδηγίας ε, περί υπηρεσιών. Τέλος, εγώ θεωρώ, λέει ένα καταναλωτή ότι είμαι Ευρωπαίος πολίτης και μπορώ και κινούμαι ελεύθερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως όταν ζητώ να αγοράσω υπηρεσίες ή αγαθά διαμεθοριακά, αισθάνομαι μεγάλη απογοήτευση, διότι εάν θέλω να πάω να αγοράσω μια υπηρεσία σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ο πολιτής μου λέει όχι, χρειάζεσαι τόπο κατοικία εδώ. Αισθάνομαι σαν να έχω μπροστά μου ένα τεχνητό σύνορο. Αυτό είναι το νόημα της ενίας αγοράς βλέπουμε από τη δήλωση αυτού του καταναλωτού ότι εδώ διακυβεύεται η ίδια αξιοπιστία της ενιαίας αγοράς. Το άνθρωπο 20 παράγραφος 2 είναι σημαντικό. Ας φροντίσουμε για την ορθή εφαρμογή του και ας βάλουμε ένα τέλος σε αυτές τις διακρίσεις. Και επόμενη διαφάνεια, σε ε, εποχές οικονομικής κρίσης η ενιαία αγορά είναι σημαντικότερη από ποτέ και αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη. Ας εκμεταλλευτούμε το δυναμικό αυτό έτσι ώστε να υποφεληθούν και οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές το μέγιστο δυνατό από την ενιαία αγορά. Και ας δούμε περισσότερα παραδείγματα αν είναι δυνατόν όπως αυτά τα χαρούμενα πρόσωπα στη φωτογραφία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σραντς. καθώς μιλούσατε για εξοικονομίες από εδώ, εξοικονομίες από εκεί, ήθελα να τις ακούσω όλες. Αλλά ε, παρακαλώ στείλτε μας ένα αντίτυπο ε, των διαφανειών ή τουλάχιστον τα αριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται και έτσι σίγουρα πολλοί θα ενδιαφερθούν. Τώρα, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μομπουάς, πρόεδρος του e-commerce Europe να ακούσουμε και τη δική του παρέμβαση για την διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, μέσα σε τρεις διαφάνειες θα σας δείξουμε περίπου ε, το δικό μας προφίλ. Η οργάνωσή μας δημιουργήθηκε πριν από ένα χρόνο με στόχο να εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις ε, που πολλούν προϊόντα και υπηρεσίες στο διαδίκτυο αλλά και διακαναλικά. Επομένως, ε, επικεντρωνόμαστε κυρίως στο διαδίκτυο, γιατί περισσότερες επιχειρήσεις θέλουν πλέον να έχουν έναν ιστότοπο. Ε, οι μεγάλες εταιρείε του λιανεμπορίου ε, καθυστερούν στην διαστηριότητά τους στο διαδίκτυο και στόχος μας είναι να προωθήσουμε αυτή τη διαδικασία στη Γαλλία μέσω του lobbying, αυτό κάνουμε και εδώ, Τώρα, ε, ε, έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα ότι έχουμε και εθνικές ε, ενώσεις που εκπροσωπούν μέσω τοπικών μελών πάνω από 4.000 επιχειρήσεις και έχουμε και 10 εταίρους, 3 επιτροπές εργασίας που απασχολούνται στα ζητήματα του καταναλωτικού δικαίου, και τη υλικοτεχνική υποστήριξη. Βλέπετε ότι τα μέλη μα προέρχονται από χώρε όπω το Βέλγιο, Ιταλία, ε, κάτω χώρε, Ισπανία και το καθεξής. Τώρα, τα καλά νέα είναι ότι ήδη υπάρχει μεγάλος κύκλος εργασιών και αυξάνεται. Ο κύκλος εργασιών μας για το 2012 ήταν περίπου 300 δις και λέω περίπου γιατί ο ορισμός ε, του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν είναι ο ίδιος με αυτό του του συμβατικού. Ε, για παράδειγμα, αν κάποιος κλείσει ένα δωμάτιο ξενοδοχείου μέσω ίντερνετ, κάποια ξενοδοχεία ε, το μετράνε ως κράτηση μέσω διαδικτύου, άλλες, άλλα ξενοδοχεία όχι. Και έτσι είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε περίπου στα στοιχεία. Όμως υπάρχει μεγάλη αύξηση, περίπου 20%. Το καλό είναι ότι η αύξηση αυτή υπάρχει σε όλες τις χώρες ακόμα και στη ΣΥΠΑ με 16% και το λέω ακόμα και εκεί γιατί ήδη είναι εξαιρετικά ε, εξελιγμένη σε αυτό το τομέα. Βλέπω λοιπόν ότι το διαδίκτυο πάει παντού. Η Ευρώπη συνολικά είναι ήδη ε, υπαριθμόν ένα αγορά στην Ευρώπη σε ό,τι φορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Όμως, είναι σαφές ότι δεν υπάρχει εσωτερική ηλεκτρονική αγορά ε, στην Ευρώπη. Αυξάνεται όμως ε, το δίκτυο 45% όχι 50% των Ευρωπαίων καταναλωτών ήδη ε, κάνουν κρατήσεις ή αγοράζουν εμπόρια και υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Από το 9% στη Βουλγαρία φτάνουμε στο 74% στη Σουηδία. Ήδη βλέπετε λοιπόν την τεράστια ανισότητα που υπάρχει στην Ευρώπη. Επομένως είναι επιτακτική ανάγκη η οικοδόμηση δικτύων ε, σε ορισμένες χώρες. Σε άλλες χώρες όπως στη Σκανδιναβία για παράδειγμα ήδη υπάρχουν αυτά τα δίκτυα. Και ήδη υπάρχει ε, αυτή η παρουσία του διαδικτύου Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, αυτή η ανάπτυξη υπάρχει παντού, σε όλες τις χώρες, ε, παρέχει καλύτερες επιλογές και καλύτερες τιμές για τους καταναλωτές. Γιατί αγοράζει κάποιος στο διαδίκτυο πρώτο τιμές, γιατί είναι και φθηνότερα τα προϊόντα, αλλά μπορεί και να τα συγκρίνει καλύτερα τις τιμές τους και δεύτερον είναι ότι είναι πολύ πιο βολικό. Μπορεί να το κάνει κανένας όποτε θέλει, στο σπίτι του, με την άνεσή του. Και τώρα πλέον και με το κινητό. Δημιουργεί θέσει εργασία. Δεν έχουμε ακόμα τα στοιχεία ε, για την Ευρώπη, αλλά περίπου 60.000 θέσει εργασία εκτιμούμε ότι συνδέονται άμεσα ή έμεσα στη Γαλλία με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και αυτό αφορά και τα δύο άκρα, αν θέλετε, και της ε, υψηλού επίπεδου και της χαμηλότερου προφίλ ε, θέση εργασία. Και μας βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη Γαλλία έγινε μια μελέτη που δείχνει ότι η μετάβαση Ε, αυτή από το να πηγαίνει δηλαδή σε ένα κατάστημα να αγοράζει στο διαδίκτυο ε, βοηθά και την προστασία του περιβάλλοντος γιατί μειώνεται μεταφορικά. Έχουμε δηλαδή απλώς τη μεταφορά του προϊόντος στο σπίτι του καταναλωτή και, δεν χρειάζεται να πάει ο καταναλωτής στο κατάστημα. Φαίνεται ότι μέχρι το 2015 το 1 τρίτο των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, θα ε, διεκπεραιώνουν στο διαδίκτυο τις πωλήσει και τι αγορέ και το 20% καταναλωτών ε, τα αγοράζουν υπηρεσίε ε, από διασυνοριακού παρόχου. Ε, Α πούμε, έχουμε το παράδειγμα του Amazon. Όταν άνοιξε το Amazon στην Ευρώπη ήταν μόνο στην Γερμανία, το Μήνο Βασίλειο και τη Γαλλία. Σε τρει χώρε. Όμω υπήρχαν πολλοί καταναλωτέ στην Ιταλία και την Ισπανία που αγόραζαν στο Amazon στους τρεις ιστοτόπους ε, των καταστημάτων. Ήταν ήδη δηλαδή διασυνοριακό από αυτή την άποψη. Πριν από δύο χρόνια άνοιξε δύο νέα καταστήματα, το ισπανικό και το ιταλικό. Δεν υπάρχει λοιπόν πλέον διασυνοριακό κατάστημα για τους Ιταλούς και Ισπανούς συναδέλφους. Αυτό, καταναλωτές συγγνώμη, αυτό δείχνει ότι πρέπει κάποιος να ικανοποιήσει τις ανάγκες ε, των καταναλωτών σε μια μεγάλη χώρα για να το κάνει αυτό ανοίγει ένα κατάστημα σε αυτή τη χώρα. Γιατί υπάρχει και το κύριο στοιχείο της γλώσσας εκεί και των προϊόντων βεβαίως. Γιατί φαντάζεστε ότι τα βιβλία δεν είναι τα ίδια στην Ισπανία και την Ιταλία. Επόμενη διαφάνεια. Θέλουμε να βοηθήσουμε τα καταστήματα αυτά να προοδεύσουν, γιατί ε, συνήθως ε, ανοίγει ένα κατάστημα σε μια χώρα και μετά παίρνουν την απόφαση να πάνε και στο εξωτερικό. Θέλουν λοιπόν την αναρμόνιση του ρυθμιστικού πλαισίου, χωρί όμως να, να υπάρχουν υπερβολικέ ρυθμίσει. Όταν ο καταναλωτής δεν είναι ικανοποιημένος, ε, έχει 15 ημέρες για να ε, δηλώσει την ε, δυσαρέσκειά του και 15 μέρες να, να επιστρέψει το προϊόν. Αλλά αν μετά από 15 μέρες το κατάστημα δεν έχει λάβει το προϊόν, τότε πρέπει παρόλα αυτά να αποζημιώσει το καταναλωτή και αυτό είναι ε, προβληματικό. Γιατί πολλές φορές αυτό θα ε, αποτρέψει τα καταστήματα της επιχειρήσεις αυτές να πάνε στο εξωτερικό. Λόγω των ε, αποστάσεων και των μεταφορικών εξόδων. Δεύτερο, ε, το δεύτερο αφορά τις πληρωμές. Γιατί σήμερα οι τρόποι πληρωμής διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ χωρών. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, έχουμε παραδόσεις και μετρητής. Δηλαδή, πληρώνονται μετρητής και παραδίδονται τα προϊόντα δεν εμπιστεύονται οι ε, να πληρώσουν κάτι, να καταβάλουν το αντίτυπο και να λάβουν το ε, προϊόν στη συνέχεια μετά μερικές μέρες. Είναι κατευθείαν λοιπόν με αντικαταβολή. Και αυτό είναι πρόβλημα βεβαίως ε, στο να πάει μια επιχείρηση στο εξωτερικό. Μετά έχουμε τα καταστήματα αναχώρα και μετά είναι η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης. Γιατί όταν, κάποιος, όταν οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν την επιχείρηση, δυσκολεύονται να την εμπιστευτούν. Στη Γαλλία το γεγονός ότι το τοπικό κατάστημα είναι γαλλικό, είναι ο βασικός λόγος που οι Γάλλοι καταναλωτές ε, το επιλέγουν. Γιατί έχουν, βλέπουν ε, ότι είναι η πενακίδα πούμε στα γαλλικά και είναι κάτι το οποίο τους εμπνέει η εμπιστοσύνη. Τελευταίο στοιχείο που θέλω να σας δείξω ε, μπορεί να μην βλέπετε τα αριθμητικά στοιχεία, αλλά βλέπετε τις διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Έχετε την ε, σύνδεση με το διαδίκτυο και μετά έχετε και τον αριθμό των ε, καταναλωτών που αγόρασαν κάτω στο διαδίκτυο. Και ο μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το, η πράσινη στήλη στη μέση. Βλέπετε αριστερά λοιπόν ότι όλοι είναι στο ίντερνετ, η χρήση είναι ήδη μεγάλη και αυξάνεται. Δεξιά όμω βλέπετε τις υπόλοιπες χώρες και εκεί θα πρέπει να, να υποδομήσουμε και δίκτυα και να βοηθήσουμε τον κόσμο ε, ε, να, να τους διευκολύνουμε να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες. Γι' αυτό και είπαμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με, αυτά τα μέτρα που ε, είναι ίδια για όλους γιατί σε αυτές τις τεράστιες ε, αγορές, την τεράστια δεκτική αγορά, τρεις ε, ε, χώρες έχουν το 50% αγοράς. Γαλλία, Γερμανία και το καθεξής. Και η Ισπανία και η Ιταλία θα πρέπει να είναι, θα πρέπει κοντά λόγω πληθυσμού, όμως υπολείπονται σε μεγάλο βαθμό. Εν ολίγης, η διαδικτυακή επιχειρηματικότητα αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν θεωρώ ότι υπάρχουν ε, φραγμοί ε, σε αυτή την ε, ανάπτυξη και θεωρώ ότι αυτά είναι πολύ καλά νέα. Ευχαριστώ. thank you very much indeed. I think for... Ευχαριστώ πολύ. Και σε πρακτικό επίπεδο πράγματι γίνεται παράλληλη δουλειά και σε άλλη Λαμέτ. Οπότε αυτό θα παρέλθουμε σε αυτό το τελευταίο και σε λίγο. τέλο. να καλωσορίσω και πάλι την κυρία Γιώχανουσαν από το Σουηδικό Σημείο Νέα επαφή Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε για τη δυνατότητα που μου δίνεται να απευθυνθώ στην Επιτροπή σας για αυτό τόσο κρίσιμο ζήτημα για την οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης και τις περαιτέρω δυνατότητες εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών και να σας παρουσιάσω την οπτική γωνία του Σουηδικού PSC εν Θα ξεκινήσω από κάτι γενικότερο, μιλώντας για την ε, σημασία της εύρυθμης λειτουργίας του PSC που για μας είναι το κριτήριο. Θέλω να πω ότι η ενιαία αγορά δεν έχει χρησιμοποιήσει πλήρως το δυναμικό που δίνει η ενιαία αγορά τη Ένωση. και εν μέρει ο τίτλο αυτού του σκέλου τη ακρόασης ε, εστιάζει στην καινοτομία. Θα πρέπει να μιλάει για καινοτομία και για άλλες εξελίξεις που αφορούν την ενιαία αγορά. Θα πρέπει μια χώρα, λοιπόν να κρατά τους ρυθμούς των εξελίξεων, να προσαρμόζεται πάντα στα νέα στοιχεία, ώστε να είναι μια σύγχρονη ενιαία αγορά. Οι υπηρεσίες παίζουν κρίσιμο ρόλο προκειμένου. Οι υπηρεσίες είναι ένα το κομμάτι κάθε παραγωγής, το έχουμε πει ξαναπεί, για όλες τις μορφές επιχειρήσεων. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του σύγχρονου εμπορίου λοιπόν οι υπηρεσίες. Ο μεταπαιδικός τομέα συνήθω δεν πολλά πλέον αγαθά πολλά πακέτο αγαθών και υπηρεσιών. Και το εμπόριο όλο και περισσότερο α, κάνει αλλαγές στον τρόπο τον οποίο παρέχει αυτές τις ε, υπηρεσίες. Και οι υπηρεσίες είναι διευκολυντές χωρίς α, τις υπηρεσίε δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το όλο εμπόριο. Θα πρέπει λοιπόν συνεχώς η αγορά να προσαρμόζεται τις νέες συνθήκες. Χρειάζονται τα κατάλληλα εργαλεία και να εδώ μπαίνω στο PSC, ε, το Point of Single Contact είναι ένα τέτοιο σημαντικό εργαλείο με το δυναμικό να βελτιώσει την ελεύθερη κυκλοφορία των ε, υπηρεσιών. Όπως βλέπετε να λέει το εθνικό μας εμπορικό μελητήριο, βλέπετε ότι ποιες είναι οι, μέσα σε πλαίσια αυτά και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και ο συντηρητικός ρόλος που έχει α, το ειδικό πίεση μαζί με άλλους δύο ακόμη φορείς. Υπάρχουν κάποιες νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία της υπηρεσίας για το πίεση. Τα απ' να βρίσκουμε τις επιχειρήσεις με ένα ενιαίο ε, web portal και να κάνουν όλες τις διοικητικές διαδικασίες online. Για να μπορεί να λειτουργεί λοιπόν το πίεση, χρειάζεται να βλέπουμε τα πράγματα από το πρίσμα των επιχειρήσεων. Άρα μια λογική της ενιαίας θηρίδας, του one-stop shop. Κάτι που πάντοτε ζητούσαν οι επιχειρήσεις. Πολύ σημαντικό σημείο κίνηση για το σουηδικό σημείο ενιαίας επαφής, το σουηδικό PSC. Βλέπετε λοιπόν σε αυτή τη διαφάνεια Βλέπετε λοιπόν πληροφορίες που πρέπει να έχουμε για τις επιχειρήσεις σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Ακούστηκε πριν ότι κάποια κρατημέλη έχουν ήδη όριμα τέτοια ε, πόρταλ. Δεν ήταν όριμο αυτό το πόρταλ ε, προκειμένο, αλλά βαστήκαμε σε υφιστάμενα στοιχεία. Βλέπετε λοιπόν ότι πήραμε υπόψη ε, την εικόνα που υπάρχει για να οικοδομήσουμε το PSC. Εδώ θα μπορέσετε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να καταλήξουμε σε μια αλυσίδα πληροφοριών και όλα αυτά στο ίδιο website. Βλέπετε με, ε, στα αγγλικά Considering Starting, Running, Developing και Closing Down. Όλα τα βήματα. Από τη στιγμή που εξετάζει και συλλαμβάνει την ιδέα μέχρι το κλείσιμο μιας επιχείρησης. Κάτω δεξιά βλέπετε το λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης EU Go που σε οδηγεί κατευθείαν ε, στο PSC. Βλέπετε ότι έχουμε αγκαλιάσει πλήρως την ιδέα ε, της, του PSC δεύτερης γενιάς που ξεπερνά και τους ίδιους τους σκοπούς της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Θέλω επίσης να πω, όπως είπε η κυρία Όμεν νωρίτερα, πόσο σημαντικό οι πληροφορίες να δίνονται σε πολλές γλώσσες. Πρέπει πέρα από την επίσημη γλώσσα της κάθε χώρας, το οποίο είναι να πληροφορίες τουλάχιστον και στα αγγλικά. Στην διαφάνεια αυτή βλέπετε ένα εξαιρετικό παράδειγμα μίας, α, ενός εντύπου... Ε, ενός Σουηδικού Δήμου που πρέπει να συμπληρωθεί. Βλέπετε λοιπόν πως είναι τυποποιημένο κείμενο στα Σουηδικά και στα Αγγλικά. Θεωρούμε ότι είναι πολύ απλό και είναι μια λύση για πολλά κρατημέλη. Λοιπόν, έχουμε καταλάβει σε κάποια κρατημέλη οι αιτήσει που είναι νομικά έγκυρες γίνονται μόνο στην επίσημη γλώσσα της χώρας. Θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι πρακτικό. Λοιπόν, αγκαλιάσαμε απόλυτα αυτή την ιδέα του PSC δεύτερης γενιάς. Αλλά θέλαμε να πάμε και παραπέρα. Ίσως να δημιουργήσουμε και το PSC τρίτης γενιάς. Θα θέλαμε λοιπόν να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτή την ιδέα για να καλύψουμε και την ιδέα της αλήθεια κυκλοφορίας αγαθών, διότι τα αγαθά και οι υπηρεσίε ε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα σήμερα και να συμπεριλάβουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο PSC. Όπως ε, ακούστηκε νωρίτερα, ένα βασικό στοιχείο του PSC είναι ο διασυνεριακός χαρακτήρας των ευρωπαϊκών διαδικασιών. Και όλες οι διατυπώσεις, ο στόχος είναι να γίνονται ηλεκτρονικά. να μπορούν να, ε, να, όλα τα τύπα ηλεκτρονικά και να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά. Μια άλλη πτυχή είναι η δυνατότητα να ε, επικυρωθεί και η ηλεκτρονική υπογραφή άλλης χώρας από το PSE. Εκεί πιστεύω ότι θα έχουμε επιτύχει και τον απότερο στόχο του PSE. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ε, δημιουργήσουμε μία λύση, μία εφαρμογή που να μην αφορά μόνο σουηδικές ηλεκτρονικές υπογραφές, αλλά και αλλοδαπές και το δοκιμάζουμε σε κάποιους δήμους. Άρα υπάρχει δυναμικό σημαντικό στο πίεση. Εγώ θα έλεγα πολύ μεγάλο δυναμικό να ε, διευκολύνουν πολύ περισσότερο τις διασυνοριακές υπηρεσίες. Και τέλος, θέλω να επισημάνω πόσο σημαντική είναι η ενημέρωση. Μιλάμε για την προσέγγιση του καταναλωτή, αλλά Χρειάζεται πληροφόρηση και των ίδιων των επιχειρήσεων. Εμείς κάναμε ήδη σεμινάρια εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των πρεσβειών. Μια σημαντική ομάδα στόχος για μας είναι η πάροχη υπηρεσιών από άλλες χώρες της Ένωσης. Και είδαμε πολύ θετική αποδοχή από αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Uh, uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί συνεχίστε να αποτελείτε καλό παράδειγμα και για τα άλλα κράτη-μέλη. Το έχουμε καταγράψει και παρατηρήσει και στο παρελθόν. Και η Άννα Μαρία το γνωρίζει αυτό. Λοιπόν, έχουμε αργήσει. Ήμουν πάρα πολύ νεκτικός μαζί σας, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα τα λεγόμενα. Θα καλέσω τους συναδέλφους να είναι πραγματικά συνοπτικοί, λακωνικοί. Φυσικά η Ανά Μαρία Κοράτσα Πίλτε θα συνοψίσει στο τέλος. Αλλά πριν από αυτό, ποια είναι τα σχόλια των συναδέλφων. Κύριε Κέπχαρτ, Στάιλερ. Ράπτη, Mr. Schmidt, no. Okay. And Mrs. Ruler, uh, Mrs. Karatza Bill, will you pick your things up at the end, whatever. Στο τέλος η συγγήτρια. Εκτός να τα ξεκινήσετε εσείς. Κυρία Κέπχαρτ, Στάιλερ, Ράπτη, με αυτή τη σειρά και μετά στους πανελίστες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις που ακούσαμε. Το σιωδικό μοντέλο πράγματι αποτελεί πρότυπο και για άλλες χώρες. Και μακάρι να γινόντουσαν τα πράγματα έτσι και στη Γερμανία ώστε να προχωρήσουμε κάπως. Είναι πραγματικά εξαιρετικό. Θα ήθελα ωστόσο να επανέλθω σε ένα πράγμα. Ευχαριστώ βεβαίως πρώτα για τις πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που κατέθεσαν οι κύριοι Σραντς και Μομπουάς και ήταν πραγματικά πολύ ανάγλυφες οι προτάσεις τους αυτές. Ωστόσο είχα την εντύπωση, και εδώ εντοπίζεται το ερώτημά μου, ότι κάπως αυτά έχουν λιγότερο να κάνουν με την ελευθερία της παροχής υπηρεσιών, με την εφαρμογή της οδηγίας δηλαδή, και περισσότερο... Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο μικρόφωνο της κυρίας Κεπχάτ. Και, και περισσότερο θα ρωτούσα εγώ πώς μπορούμε να φροντίσουμε ώστε οι προσφορές που γίνονται από πλευράς ορισμένων ε, παρόχων υπηρεσιών να γίνονται πραγματικά προς όλους τους πολίτες και όχι επιλεκτικά προς ορισμένους εκάστοτε. Κοιτάξτε, εδώ είναι θέμα πολιτικής ανταγωνισμού. Άλλος νομοθετικός τομέας που πρέπει να εξεταστεί. Η κυρία Στάιλερ. Κάτι παρόμοιο. Πάλι πολιτική ανταγωνισμού. Επειδή κάποιος μίλησε για το Amazon που ελέγχεται τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο διότι ασκεί φόρο αποφυγή. Δεν είναι, απόλυτα παράνομη, δεν είναι βέβαια η φόρο αποφυγή. Εάν λοιπόν έχουν κέντρα διανομής και αυτά τα κέντρα διανομής και πάντως στην περίπτωση της δικής μου χώρας αν έχει λάβει κρατικές επιχορηγήσεις μπαίνει ένα θέμα φορολογίας Χρειάζεται λοιπόν κάποια διερεύνηση. Θα ήθελα κάποιες σκέψεις σας πάνω σε αυτό γιατί όπως ξέρετε υπάρχει και το θέμα της λεγόμενης high street και του τι γίνεται δηλαδή στα καταστήματα και αρχίζουν σιγά σιγά οι άνθρωποι να αμφισβητούν λίγο γιατί λένε ναι μεν θέλουμε υπηρεσίες, τα θέλουμε όλα αυτά τα πράγματα και ορισμένες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και στο ηλεκτρονικό εμπόριο και βέβαια διατηρούν και καταστήματα στο λεγόμενο high street. Αλλά βέβαια μπαίνουν πάλι κάποια θέματα φορολογία κλπ. Θα ήθελα να ακούσω κάποιε σκέψει. σα. Αυτό είναι στην πραγματικότητα υλικό για μια ακόμα ακρόαση. Κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, φέρνω στο μυαλό μου την οδηγία για την προστασία των καταναλωτών και θυμάμαι ότι τότε το κύριο διακύβευμα ήταν το επίπεδο εναρμόνισης. με εναρμόνιση ή μίνιμουμ εναρμόνιση. Το ερώτημά μου είναι ε, κυρίως προς τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών εάν εκτιμά ότι η πρόβλεψη της Επιτροπής για με εναρμόνιση θα βοηθήσει τελικά τους καταναλωτές ή όχι και σε τι βαθμό. Ευχαριστώ. Um, anybody else? Άλλος κανείς, παρακαλώ. Τότε. Ας ακούσουμε πρώτα την κυρία Γιώχανσον, μετά τον κύριο Μομποάση και μετά Σραντς. Δεν απευθύνθηκαν ειδικά σε μένα οι ερωτήσεις, αλλά για, τις πρώτες, για την πρώτη μάλλον ερώτηση α υπενθυμίσω την, ε, τα, τα τα κέντρα Solvit που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και εμείς έχουμε το, ε, στο, στο κέντρο μας έχουμε ε, τέτοιο Solvit. Και τα έχετε ενσωματώσει αυτά. Α, μάλιστα, ναι. Μουμπουάς. Amazon και φορολογικά. Το ίδιο, η ε, ίδια κίνηση υπάρχει στη Γαλλία. Αυτό που λέμε εμείς, η French Trade Association, είναι ότι το φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι δίκαιο. Και όλες οι εταιρείε που δραστηριοποιούνται στη Γαλλία πρέπει να έχουν ε, να υφίσταται την διαφορολογία και το 99,9% των, των μελών μου διασαρεστούνται με την Amazon. Η Amazon βέβαια είναι πανέξυπνη και παίρνει επιδοτήσεις για τα κέντρα διανομής, κάνει και κάποιο ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων πόλεων γιατί δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτό όμως ωστόσο δεν είναι παράνομο. Πάντως στο Βρετανικό Κοινοβούλιο τέθηκε το θέμα των εφιών αυτών στρατηγίων που έχει βάλει και η Γιβραλτάρ, Λουξεμβούργο κλπ. Είναι κάτι όμως που μπορείτε να περάσετε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί ο κόσμος έχει αντιληφθεί τι γίνεται και δεν είναι ικανοποιημένος. Θα είδατε ίσως και μια κοινή επιστολή Μοσκοβισής Άμπικος Μπόρν στους Financial Times για το θέμα αυτό. Για το ότι δηλαδή οι πολυεθνικές θα πρέπει να πληρώνουν φόρους. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Ένα πράγμα που με εξέπληξε πολύ δυσάρεστα στο G8 όπου ο Ερικ Σμιτ μαζί με την Κριστίν Λαγκάρντ που ήταν ακόμα τότε Γαλλίδα Υπουργό ε, Οικονομίας και είπε τότε εμείς να φτιάχνουμε την οικονομία, εσείς να φτιάχνετε τα δίκτυα. Και ε, για τους, για τους μεγάλους αυτούς ε, ε, οργανισμούς, Google, Amazon κλπ. Τώρα για την προσφορά συνήθως τα καταστήματα προς κάνουν τη μεγαλύτερη προσφορά στους καταναλωτές. Φνακ είναι γνωστή, η Φνακ που ε, πουλάει δίσκους, βιβλία κλπ. Έχουμε, έχει και ηλεκτρονικό εμπόριο και για παράδειγμα και στους Ιταλούς και για παράδειγμα τα Ιταλικά βιβλία πάνε στην Ιταλία, τα γαλλικά στη Γαλλία και μεταφέρονται από εκεί. Εκτός εάν υπάρξουν περιορισμοί όπως με συνδρομές στο ίντερνετ όπου η προσφορά είναι πολύ τοπική, περιορισμένη τοπικά δηλαδή όπως για τηλεόραση κλπ. Και η δεύτερη ερώτηση δεν δε θυμούμαι ποια ήταν η τρίτη, α ναι, εναρμόνιση. Λέχθηκε ότι για την προστασία των καταναλωτών είναι πλήρους εναρμόνισης και αυτό το έχει αποφασίσει και το Κοινοβούλιο. Α, όχι σε όλους τους τομείς όμως. Αλλά για internet business ναι. Και εμείς θεωρούμε ότι είναι μεγάλη βελτίωση. Αλλά βέβαια θα τα συζητήσουμε και αύριο αυτά με την κυρία Κέπχαρτ. Α, δεν θέλουμε να βάλουμε οπωσδήποτε και ένα κοινό ευρωπαϊκό νόμο πωλήσεων. Κύριε Σράντς, ήσασταν πραγματικά το αστέρι του σημερινού απογεύματος και πολύ ευχαρίστω σας δίνω τον τελικό λόγο. Πριν ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Μπίλτ, οι υποθέσεις που σας παρουσίασα είναι του πεδίου εφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 Εκεί ήταν πάντοτε η διαφορά των τιμών. Όταν ο καταναλωτής ζητεί προσφορά υπηρεσίας και όταν επιλέγει τη φθηνότερη τιμή, τη χαμηλότερη τιμή δηλαδή, του αρνούνται την προσφορά αυτή της υπηρεσίας, αυτές είναι οι υποθέσεις οι οποίες εμπίπτουν στο 20 παράγραφος 2. Συν το χρόνο, νομίζω θα έχουμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, γιατί οι καταναλωτές κοιτούν στο διαδίκτυο, ψάχνουν να βρουν διαφορετικές προσφορές και όταν βρίσκουν ευνοϊκότερες τιμές σε άλλες χώρες βέβαια θέλουν να τις ε, χρησιμοποιήσουν, θέλουν να τις ε, εκμεταλλευτούν. Στο μέλλον λοιπόν θα έχουμε περισσότερες τέτοιες ε, υποθέσεις και είναι σημαντικές διότι οι καταναλωτές απογοητεύονται, χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην ενιαία αγορά και αυτό πρέπει κάπως να το αντιμετωπίζουμε. Ένα άλλο θέμα που δεν μίλησα πολύ στην παρέμβασή μου είναι εάν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι, τότε έχει καλός. Έχει καλός η άρνηση της προσφοράς υπηρεσίας. Και τότε και εφόσον συμφωνούν και οι, οργανώσει οι οργανώσεις προστασίας καταναλωτών. Αλλά όπως είπα, σύν το χρόνο, ορισμένοι από αυτούς τους αντικειμενικούς λόγους θα πάψουν να ισχύουν. Όπως είπε κάποιος προηγουμένως, η νέα οδηγία προστασίας καταναλωτών, που ελπίζω ότι θα εναρμονίσει την, το δίκαιο προστασίας καταναλωτών και στο μέλλον, όπως είπα, καθώς θα περνά ο χρόνος, θα αρθεί το εμπόδιο αυτό. Και ένα άλλο ε, εμπόδιο είναι η ανάκτηση των χρεών διότι οι ε, έμποροι δεν θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλες χώρες γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν τα λεφτά τους τελικά. Εγώ στο, στη δουλειά μου χρησιμοποιώ καθημερινά το European Repayment Order και λέω και στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν αυτήν την ε, ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής για να εισπράξουν χρήματα τα οποία δεν τους έχουν αποδοθεί. Όπως είπα λοιπόν, καθώς θα περνά ο χρόνος θα δούμε ότι θα έρονται τέτοια εμπόδια και θα προχωρούμε περισσότερο σε εφαρμογή πολιτικών ενιαίας αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στη συνάδελφο κυρία Μπίλτς για να απαντήσει. Σίγουρα θα είναι πολύ σύντομες και περιεκτικές αλλά και ενδιαφέρουσες ε, οι παρατηρήσεις σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και την Βρυγκίτ και τη Διαρία από τη Γραμματεία και τους συναδέλφους σας, γιατί πραγματικά το πάνελ σήμερα το απόγευμα ήταν φανταστικό. Αντλώ έμπνευση και πολύ σημαντικά συγκεκριμένα συμπεράσματα. Και πραγματικά ε, θέλω να παραμείνω σε επαφή μαζί σας, ε, παραμείνετε κι εσεί σε επαφή μαζί μα να μα ενημερώνετε και το καθεξή. Βλέπω λοιπόν τη σημερινή συζήτηση ότι συμφωνούμε ότι χρειάζεται λιγότερο κατακαιρματισμό, μεγαλύτερη εναρμόνιση, μία ανοχή στη μη υλοποίηση οδηγία περιπηρεσιών και ότι πρέπει να επικεντρωθούμε πραγματικά στην ε, βελτίωση της ε, υφιστάμενης κατάσταση. Δεν χρειάζεται να επανεφεύρουμε τον τροχό. Είδα λοιπόν ότι υπάρχει μια διαφωνία σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή. Πολλοί αναφέρθηκαν σε ζητήματα πέραν του αντικειμένου ε, τη οδηγία, σε άλλε οδηγίε και το καθεξής. Παράλληλα, στην ψηφιακή Ευρώπη πρέπει να έχουμε κατά νου την αλληλεπίδραση. Όταν δηλαδή υλοποιούμε, εφαρμόζουμε την οδηγία υπηρεσιών, την αλληλεπίδρασή τη, λοιπόν με άλλε ε, ε και σε τη αφορά και την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Ε, Δυστυχώ δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των κρατών μέλων εδώ και η Ιρλανδική Προεδρία δεν έκανε τον κόπο να παραμείνει. Και ενώ αναφέρθηκε ότι είναι τόσο σημαντική αυτή η ακρόαση ε, για τους καταναλωτές, δεν μπήκαν καν στον κόπο να ακούσουν την άποψη των καταναλωτών γιατί αυτή είναι η ομάδα που μας απασχολεί. Έχουμε μια ευθύνη εδώ λοιπόν. Αυτή, αυτό το έργο να μην αποτελέσει αντικείμενο διχασμού, ιδεολογικού διχασμού μεταξύ αριστεράς, δεξιάς, ε, σωματείων και ε, εργοδοτών. Όταν κάποιο έχει θέση εργασία, ε, οι συνθήκε εργασία δεν έχουν σημασία γιατί κάποιο έχει μια δουλειά. Και έτσι είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε Θέσει εργασία με αυτή την οδηγία. Και οποιοδήποτε συμφωνεί μαζί μου μπορεί να συνεργαστεί μαζί μου. Έχουμε δυόμιση σελίδε. Ξέρετε πώ πάνε τα πράγματα στο Κοινοβούλιο, δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα. Έτσι συμβαίνουν τα πράγματα στο Κοινοβούλιο. Σε κάθε ψήφισμα θέλουμε να ε, τα λύσουμε όλα, αρχίζουμε να πλατιάζουμε. Εγώ δεν πρόκειται να το κάνω αυτό. η δική μου πολιτική ομάδα, το ΕΛΚ, θα είναι ενωμένη σε ό,τι αφορά το αντικείμενο το πεδίο εφαρμογή. Θα είμαστε σοβαροί απέναντι στο ζήτημα των θέσεων εργασία στην Ευρώπη. Βεβαίω και πρέπει να εξισορροπήσουμε την κοινωνική διάσταση, κύριε Σφόρτ. Βεβαίω και είναι σημαντικό. Έχουμε εθνικού νόμου, συλλογικέ συμβάσει στι πατρίδε μα. Κάποιο ανέφερε ότι δεν υπάρχει καν κατώτατος μισθό σε όλα τα κρατη Και θα ήθελα να παραθέσω το άρθρο 1 της Οδηγίας Περιπηρεσιών. Η οδηγία δεν επηρεάζει το εργατικό δίκαιο ή τι συμβατικέ διατάξει, ό,τι φορά τι εργασιακές συνθήκες, συνθήκε απασχόλησης και τη σχέση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Ε, η κυρία Νίλσον που εκπροσωπεί τα σωματεία της Ευρώπης είπε εδώ ότι συμφωνεί ότι δεν θα ξανανοίξουμε αυτή την οδηγία και συμφωνώ. Θα την τραβήξουμε ούτως ώστε να καλύπτει και τις ψηφιακές υπηρεσίες που δεν υπήρχαν το 2006. Θα γίνει λοιπόν πιο ελαστική αυτή η οδηγία για να καλύψει αυτά τα νέα στοιχεία θα ανταποκριθούμε στους ε, νέους ε, τρόπους ε, με τους οποίους θέλουν να ζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Δεν θα ξεκινήσουμε εκ νέου αυτή την νομοθετική διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα με τις κοινέ μας προσπάθειες, ούτως ώστε να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι δεν είναι αρκετό να έρχονται εδώ και να, ακούσουμε, να, ακούμε, να έρχονται εκείνοι εδώ να μας λένε τα ίδια που μας λένε και οι εμπειρογνώμονες να μας πούνε δηλαδή ότι πρέπει να υλοποιήσουμε την οδηγία χωρίς να μας πούνε τι κάνουν οι ίδιοι, ε, τι ακριβώς κάνουν για την υλοποίηση. Θέλουμε απαντήσεις, όχι αναλύσεις από εκείνους. Αναλύσεις κάνουν και άλλοι. Όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό ως δικαιολογία για να καθυστερήσουν και να αναβάλουν την υλοποίηση όσων μπορούν να υλοποιηθούν σήμερα. Και αναφέρθηκαν αρκετά τέτοια παραδείγματα που μιλούν από μόνα τους. Κλείνοντας, έχω πολλά να πω και ζητώ συγγνώμη που δεν είμαι σε θέση να τα συνθέσω όλα καλύτερα. Όμως θα διαβεβαιώ όλους ότι σας ακούσαμε με προσοχή, σημειώσαμε τις παρατηρήσεις σας, θα αναλύσουμε τα όσα είπατε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Well, thank you very much indeed. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα Μαρία. Και βεβαίως ε, ευχαριστούμε και την ομάδα σου και τους Χιώδη. Θα μας στείλει ε, την έκθεση προς μετάφραση ε, 15. Την περιμένουμε λοιπόν. Θα την εξετάσουμε στις 24-25 Απριλίου. Θα περάσουμε καλά σίγουρα. Και η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η 7 Μαΐου. Και θα δούμε μετά το επόμενο χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ και πάλι τους αναπομείναντες ομιλητές. Βεβαίως ευχαριστούμε και τους προηγούμενους που έφυγαν. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους ε, που ε, ήρθαν εδώ μαζί μας. Τέλος να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε και νέο ενημερωτικό φυλάδιο. Αν θέλετε μπορείτε να συμπληρώσετε στοιχεία σας για να το λάβετε. Κλείνει λοιπόν ε, το ανοιχτό επίσημο τμήμα της συνεδρίασής μας. Αύριο το πρωί στις 9 συνεχίζουμε και η συνάντηση των συντονιστών θα ξεκινήσει το στομότερο δυνατόν. Παρακαλώ οι υπόλοιποι να αποχωρήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα γιατί η συνεδρίαση θα γίνει για κλεισμένο των θυρών.